Hello, good afternoon to everybody. Καλησπέρα σε όλους. Ριπρεντιάμο. Να συνεχίσουμε τις εργασίες μας σε αυτό το τόσο σημαντικό σεμινάριο με την έναρξη του δεύτερου πάνελ για την πρόθεση της συμμετοχής των πολιτών. Ε, η πρωινή συζήτηση ήταν μια συζήτηση ιδιαίτερα έντονη και έφερε στην επιφάνεια τις ε, πάμπολες περιπτώσεις, ε, αρκετές φορές αδικαιολόγητες ε, προσκομμάτων που εμφανίζονται σε σχέση με τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Κυρίως όλα όσα αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πολιτών, τα θέματα της γραφειοκρατίας, το, την έλλειψη αμοιβαιότητα, την έλλειψη πληροφοριών και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαμε και άμεση εμπειρία και στήριξη της Επιτροπής Αναφορών η οποία αδιαμφισβήτητα είναι ε, προνομιούχος αυτή την περίπτωση. Το 2012 μόνον λάβαμε πάνω από 2.300 αναφορές. Το μέσο της αναφοράς είναι κάτι το οποίο απορρέει από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, αναγνωρίζεται στη συνθήκη και κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να αποτανθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να καταγγείλει την ε, ε, λανθασμένη ή την ε, απουσία εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου από πλευράς τοπικών και εθνικών αρχών ή να συνεισφέρει και στην θεσμική συζήτηση και στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο της Προεδρίας μου, διότι βρίσκομαι πλέον στο τέλος του τέταρτου έτους Προεδρίας, εκτίμησα τις μεγάλες δυνατότητες που μας προσφέρει αυτό το μέσο, το οποίο πολύ συχνά αποκάλυψε πολύ σοβαρές παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. Κατορθώσαμε αρκετές φορές μέσω σημαντικών αναφορών να επισέλθουμε και στην ε, νομοθετική συζήτηση όπως συνέβη για παράδειγμα με την ε, πολύ γνωστή περίπτωση της Συμφωνίας Άκτα, όπως έγινε και προσφάτως με την ε, Συμφωνία για την Αλία. Και στις δύο περιπτώσεις ως Επιτροπή Αναφορών ε, είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών για το θέμα που σχετίζεται με την Άκτα, περίπου 2 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών εξέφρασαν την ανησυχία τους ε, στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τώρα την πολιτική αλληλείας, έχουμε περίπου 900.000 πολίτες ε, οι οποίοι απευθύνθηκαν σε μας διότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης θα έπρεπε να δράσει λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα καταγγέλουν οι πολίτες. Αυτό βεβαίως δεν ε, σημαίνει ότι το δίκαιο που μας εγγυούνται οι συνθήκες ε, δεν ε, ε, μπορούν να το ασκήσουν και οι πολίτες τους. Ο κάθε πολίτης μπορεί μεμονωμένα να απευθυνθεί στην Επιτροπή Αναφορών για τα θέματα τα οποία τον αφορούν και μπορεί να συνεργαστεί για την καλύτερη χρήση του μέσου της ευρωπαϊκής συμμετοχής. Έγιναν αρκετές προσπάθειες οι οποίες ε, μεταφέρθηκαν ε, στις ε, συνθήκες για να δώσουμε νέες δυνατότητες στην συμμετοχή των πολιτών σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Με την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Αμβώνες αναγνωρίστηκε και η δεσμευτική ισχύ της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και έχει εισαχθεί και η διαδικασία συναπόφασης μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 90% των θεμάτων της ε, ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και έτσι διασφαλίζεται η μεγαλύτερη συμμετοχή, η μεγαλύτερη δημοκρατική συμμετοχή στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων και μεταξύ άλλων έχει συμπεριληφθεί και μια εξαιρετική καινοτομία της δυνατότητας πρωτοβουλίας, νομοθετικής πρωτοβουλίας των πολιτών. Για πρώτη φορά λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα ένα εκατομμύριο πολίτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη να προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα νομοθεσία. Η Επιτροπή Αναφορών ε, συμμετέχει άμεσα σε αυτή τη διαδικασία ε, διότι πρέπει να εγκρίνει τις πρωτοβουλίες που προτείνουν οι πολίτες. Ε, συμμετείχαμε στην έγκριση του, ε, του κανονισμού 211-2011, ε, ο οποίος ρυθμίζει τη διαδικασία για την πρωτοβουλία των πολιτών και η Επιτροπή μας θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία όταν θα γίνεται η ακρόαση των πολιτών που προηγείται της διαδικασίας ε, έγκρισης της οδηγίας ε, που έχουν κάνει οι πολίτες, ε, τις νομοθεσίες που έχουν κάνει οι πολίτες. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τελευταίες πρωτοβουλίες των πολιτών που έχουν καταγραφεί, που είναι ακόμα στη διαδικασία συλλογής υπογραφών, αφορούν το θέμα της πολιτικής συμμετοχής. Ένα θέμα στο οποίο θα σταθεί το επόμενο πάνελ. Και η πρωτοβουλία των πολιτών με τίτλο Let Me Vote αφορά το δικαίωμα των πολιτών να ψηφίζουν στο κράτος μέλος σε όλε τι εκλογικέ αναμεκτρήσεις με ε, ίσους όρου, επίση όρους με τους ε, πολίτες ε, του κράτου μέλου. Θέλει να επιλύσει και το πρόβλημα του δικαιώματος ψήφου το οποίο στερούνται αρκετοί πολίτες που μένουν μόνιμα σε κράτη-μέλη τα οποία δεν είναι τα κράτη-μέλη καταγωγής τους. Πρόκειται για ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν συχνότερα οι πολίτες από ό,τι είδαμε από τις αναφορές που απευθύνονται στην Επιτροπή μας. Και ε, το πρόβλημα αυτό ε, φέρνει στην επιφάνεια ένα πολύ σημαντικό βραχικύκλωμα, διότι δεν μπορούμε αφενός ε, να προωθούμε την ελευθερία κυκλοφορίας και αφετέρου να αγνοούμε πολύ σοβαρές συνέπειες, όπως για παράδειγμα τη στέρηση του δικαιώματος ψήφους, για να μην σταθώ και στα υπόλοιπα, και ε, να μην αναλαμβάνουμε και να βρούμε κατάλληλες λύσεις για το θέμα αυτό. Προσφάτως, στη χώρα μου, στην Ιταλία, ε, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πόσες ελλείψεις έχει το σύστημά μας ε, διότι ήταν πάρα πολλοί οι νέοι οι οποίοι ε, αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε προγράμματα ερέσμους σε όλη την Ευρώπη και οι νέοι αυτοί υποχρεώθηκαν να μην ψηφίσουν εκτός και αν αναλάβουν οι ίδιοι τα έξοδα για να επιστρέψουν στη χώρα τους και να ψηφίσουν και να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους. Επίσης, αργότερα θα είναι πολύ σημαντική και η μαρτυρία που θα ακούσουμε μιας Αγγλίδας συμπολίτησή μας, η οποία υπογράφει μια αναφορά και καταγγέλει ε, κάποια πρακτικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου της και αυτό σε συνέπεια μιας απόφασης ε, την οποία θα έπρεπε να υποστηρίξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μεταφέρει την ε, διαμονή της εδώ και χρόνια, τον τόπο μόνιμης διαμονής της ε, στην Ισπανία και αυτό τη στέρισε το θεμελιώδης δικαίωμα ψήφου της. Όσον αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας, η ελευθερία κυκλοφορίας είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς όταν αναρωτιόμαστε τι ακριβώς ε, περιλαμβάνει αυτό το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να το συνδέουμε και με αυτό το πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωμα ψήφου είναι θεμελιώδες και είναι και θεμελιώδης απόδειξη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών ε, στην ζωή της χώρας τους και θα πρέπει σαφώς να κάνουμε ε, ακόμα περισσότερες προσπάθειες φέτος το, ε, που είναι η χρονιά η οποία είναι αφιερωμένη στους πολίτες και θα πρέπει στη διάρκεια αυτού του έτους να προσπαθήσουμε να άρουμε τα φραγμούς που αποτελούν ανάχωμα στην άσκηση αυτού του δικαιώματος. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε την ε, σύντομη παρέμβασή μου για να δώσω το λόγο ε, στον συνάδελφο, ε, στον δήμαρχο Γιώργη Γεμέζη, που είναι δήμαρχος της πόλης Γκοντέλου στην Ουγγαρία, εισηγητής από την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και τα δικαιώματα ψήφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του εισηγητή, ο οποίος τονίζει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή σε τοπικές και δημοτικές εκλογές των πολιτών, ε, που είναι ε, υπήκοοι άλλη χώρα μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διαμένουν μόνιμα σε άλλη χώρα και αυτό είναι να πάει προ το τμήμα τη Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Θα είναι ιδιαίτερη χαρά λοιπόν να ακούσουμε την ε, παρέμβασή του. Ε, εύχομαι σε όλου να είναι πολύ καρποφόρα η συγκεκριμένη ημέρα και ελπίζω να βρούμε χρήσιμους τρόπους για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύσεις και να μην γεμίσουμε απλώς την ημέρα μας με θεωρίες που δεν θα γίνουν ποτέ πράξη. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Με μεγάλη χαρά συμμετέχω σήμερα σε αυτή την ακρόαση όπου θα ανταλλάξουμε απόψεις για την τοπική και περιφερειακή επίπτωση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Τα θέματα αυτά έχουν καθημερινή επίπτωση στη καθημερινή ζωή των πολιτών μας και ο, το καλύτερο μέρος για να ε, συζητήσουμε αυτά τα θέματα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικοί μας ε, τοπικά και περιφερειακά βλέπουν κάθε μέρα την απογοήτευση και την ε, αγανάκτηση των πολιτών μας, ε, οι οποίοι καθημερινά αντιμετωπίζουν την μεγάλη οικονομική κρίση. Οι σπιγομετρήσεις της κοινή γνώμης δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ε, σε οικονομική κρίση, αλλά πάσχει και από μια κρίση εμπιστοσύνης. Αυτή η δημόσια δυσπιστία δεν είναι κάτι το καινούριο και πρέπει να επανικοδομήσουμε ε, αυτή την εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αλλά είναι δύσκολο. Ο Ζακ Ντελόρ είπε πριν από πολλά χρόνια ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή κοινή αγορά και ότι δεν είναι εύκολο να ερωτευθεί κανείς τα τους όρους της ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική αγορά κλπ. Επαναλαμβάνω ότι συμφωνώ με αυτό, αλλά ε, η εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι δεδομένου ότι υπάρχει ένα πλήρες κοινοβούλιο να αντιπροσωπεύει ισότιμα και πλήρως τους Ευρωπαίους πολίτες σε όλα τα θεσμικά όργανα. Και πρωτοβουλίες όπως Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πολύ μεγάλη επιρροή. Χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία, περισσότερη συνεργασία. Ίσως να μην έχουμε αντιληφθεί πλήρως το τεράστιο έργο που έχουμε μπροστά μας επί καθημερινής βάσεως. Είμαι πεπισμένος ότι έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να γράψουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών και ουσιαστική ε, ο ουσιαστικός σύνδεσμος ε, για όλα αυτά είναι η Ευρωπαϊκή εισαγένεια. Η Ευρωπαϊκή Ισαγένεια είναι μια παράλληλη έννοια με την εθνική υπηκότητα, την εθνική Ισαγένεια και επίσης συμβαδίζει και με την ε, τοπική ιδιότητα και τα τοπικά χαρακτηριστικά. Ε, ε, όπως είπαμε. Λοιπόν, συμβαδίζει αυτή η σαγένεια με ένα μεγάλο πακέτο, μια δέσμη δικαιωμάτων, τα οποία έχουν παγιωθεί ε, στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ισαγένεια είναι μια χειροπιαστή έννοια η οποία προσδίδει όλα, όλες τις απαραίτητες ιδιότητες στον Ευρωπαίο πολίτη και ξεπερνάει το συμβολισμό. Μία ευρωπαϊκή εισαγένεια δείχνει ε, την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης για κάθε μας πολίτη. Και ε, πρέπει συνέχεια να επαναλαμβάνουμε ότι η, εθνική, η ευρωπαϊκή εισαγένεια προάχει τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλουμε όλες μας τις προσπάθειες και στο τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας που συζητήθηκε το πρωί ε, καθιστά πραγματική την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διάσταση δηλαδή της Ένωσης, με βεβαίως το σεβασμό της ε, ποικιλομορφίας. Ε, πρέπει τα δικαιώματα αυτά ε, να ωφελούν όλους τους πολίτες τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα όπως τα δικαιώματα υποβολής αναφορών. Ε, πρέπει να χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα για να καταπολεμήσουν τις διαφαινόμενες τάσεις αντιδημοκρατικής Ευρώπης ανεξάρτητα από την υπηκότητά τους, τη γλώσσα τους, τους πολιτιστικούς τους δεσμούς και την εθνότητά τους, οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν την πρώτη και την τελευταία λέξη στη διαμόρφωση της, ε, του νομικού πλαισίου. Και είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα, όλες οι ενώσεις, όλες οι πλατφόρμες που υπάρχουν ε, διασυνοριακά οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στο να διαδώσουν και να ενημερώσουν τους πολίτες τα δικαιώματά τους. Πρέπει να βρουν τα μέσα να καταπολεμήσουν πολλά εμπόδια τα οποία υπάρχουν στην άσκηση των δικαιωμάτων που ανακύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια στην έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια του 2010, οι οποίες, πτυχές τις οποίες συζητήθηκαν το πρωί, αναφέρονται οι προτεραιότητες της Ιθαγένειας. Πρώτη και κυριότερη είναι η ε, υλοποίηση των δικαιωμάτων και η εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και τα δικαιώματα έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα στους καταστατικούς χάρτες των κρατών μελών. Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν στο γράμμα του νόμου, αλλά πρέπει να τις μετατρέψουμε και σε πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να εξασκήσουμε περισσότερη πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις να ε, διαφυλάξουν αυτήν την ε, ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να αποφύγουν και να ξεπεράσουν ε, άχρηστα γραφειοκρατικά εμπόδια και προσκόμματα, τα οποία τους δυσκολεύουν τη ζωή. Αυτό ε, πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα όταν καλωσορίζουμε νεοεισερχόμενους Ευρωπαίους πολίτες. Επίση, είναι ευθύνη μας να συνοδεύουμε Ευρωπαίους πολίτες όταν ε, χρειάζονται τη βοήθειά μας για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Έτσι ώστε να είναι συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι πολίτες και να αναγνωρίζουν, να ξέρουν ακριβώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό ακριβώς η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, είναι ε, το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών ε, και εμείς έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να τους βοηθήσουμε. Εμείς ως πολιτικοί αλλά και ως τοπικοί εκπρόσωποι και στελέχοι της διοίκησης πρέπει να παράσχουμε αυτές τις, ε, αυτή τη βοήθεια αυτή την, και την πληροφόρηση το Ευρωπαϊκό Έτος της εισαγένειας ε, είναι μια πολύ κατάλληλη ευκαιρία συζήτηση αυτών των θεμάτων ένα χρόνο πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα γίνει του χρόνου. Πιστεύουμε ε, ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται, οικοδομείται ε, ο Ευρωπαϊκός Δήμος, με την έννοια δηλαδή την αρχαία, ο Δήμος, η κοινότητα της Ευρώπης η οποία είναι βεβαίως ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα. Η ευρωπαϊκή γίνει. Είναι το ζωτικός ε, κόμβος επικοινωνίας, ο κομβικός σύνδεσμος ε, μεταξύ των πολιτών και των διοικήσεων ε, και μόνο μία συνειδητοποιημένη ευρωπαϊκή ε, ταυτότητα μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη τοπικά και περιφερειακά. Το 2010, η ονομοσία του 2013 ως έτους Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας δείχνει ότι υπάρχει ζωτικότατο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και την και πολλές διευκρινήσεις ε, πτυχών που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ισαγένεια και που δεν τις ξέρουν οι πολίτες μας. Το όπως, όπως χρειάστηκαν χρόνια να καθιερωθεί το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο, το οποίο βοηθά βεβαίω ε, στην εδραίωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, έτσι πρέπει και εμείς να προσέξουμε τώρα ε, να προβάλλουμε όσο δυνατόν καλύτερα το έτος αυτό. Ε, και θα υιοθετηθούν ε, φέτος δύο οδηγίες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Πιστεύω ότι η επικύρωση, η υιοθέτηση αυτών των δύο οδηγιών θα βοηθήσει να προάγει αυτό το θέμα. Η προαγωγή των ε, εκλογικών δικαιωμάτων είναι και ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε. Αυτό περιέχεται στη μία πρόταση οδηγίας και ζητάει από την Κομισιόν να αναλάβει δράση για να ενσαρρύνουν τα κράτη-μέλη ότι αυτά τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα ψήφου ε, ε, είναι εγγυημένα σε όλους τους πολίτες. Και να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη ε, να βοηθήσουν τους πολίτες, να διευκολύνουν μάλλον τους πολίτες την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, του εκλογικού καθήκοντος. Όχι μόνο στις τοπικές εκλογές, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Και γι' αυτό υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας Let Me Vote. Άφησε με να ψηφίσω. Και έχουμε διατυπώσει πολλά, μέσα, πολλά μέτρα συγγνώμη, τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν ε, στην άσκηση του δικαιώματος αυτού. Τελικά θα υποβληθεί μία πρόταση κανονισμού για την χρηματοδότηση ε, του Ευρωπαϊκού Φορέως ε, για τον πολίτη και για την ενίσχυση όλων των, μέσων αυτών που αφορούν τοπικές και περιφερειακές αρχές. Πιστεύω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της συνδυτοποίησης ευρωπαϊκών πολιτικών και να γεφυρώσουν τις, ε, την τοπική, περιφερειακή και εθνική ζωή των πολιτών κάθε ευκαιρία ανοιχτή συζήτηση ευρωπαϊκών θεμάτων πρέπει να την ενθαρρύνουμε και επίσης πρέπει να ενθαρρύνουμε την ε, συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Με την ευκαιρία αυτή ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όλους τους εταίρους και ενδιαφερόμενους να αναλάβουν υπεύθυνα το ρόλο τους, να εξασκήσουν τις ευθύνες τους και να επιτύχουν, να σημειώσουν επιτυχία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους προάγοντας την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Όχι μόνο στις εκστρατείες ενημέρωσης και όχι μόνο το 2013. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ε, που θα καθορίζει όλες τις μελλοντικές πολιτικές στην καθημερινή μας ζωή. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι και συναισθηματικό το θέμα αυτό. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ενισχύσουμε δραστηριότητες των πολιτών, δραστηριότητες ε, και πρωτοβουλίες ε, της κοινωνίας των πολιτών, ε, εκδηλώσεις δημόσιες και οτιδήποτε προάγει την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Επίσης θέλω να αναφέρω ε, στους συναδέλφους ότι υπάρχουν και πολλά, πολλοί άλλοι φορείς, οργανισμοί, Ινστιτούτα που εκτελούν παρόμοιες εργασίες. Και ανα πάσα στιγμή πρέπει να έχουν κατά νου την περιφερειακή συμμετοχή και να λαμβάνουν υπόψη στην εκπώνηση της πολιτικής και της στρατηγικής τους ε, το τοπικό και περιφερειακό δημοκρατικό στοιχείο. Διαφορετικά δεν, ε, δεν εννοείται ευρωπαϊκή πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι εμπλεκόμενες και ενδιαφερόμενες αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να ε, τονίσουν την ευρωπαϊκή εισαγένεια. Γιατί έτσι θα προσθεθεί και περισσότερη αξία, περισσότερος δυναμισμός, περισσότερο δημοκρατικό στοιχείο στη ζωή των πολιτών μας. Και τέλος, αυτό είναι... And all of them. EU is not μία παράκληση, μία έκκληση σε όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κατάστημα που πάμε να ψωνίζουμε αυτά που μας ενδιαφέρουν και μας αρέσουν. Είναι μία, ε, ένα οικοδόμημα, μία μηχανή δράσης, ένας μηχανισμός δραστήριος και πρέπει να, στο οικοδόμημα αυτό να αισθάνονται όλοι σαν το σπίτι, σπίτι τους. Όλοι όσοι είσαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να αισθάνεστε Ευρωπαίοι. Όπου και να είστε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you to you, miss. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γκέμεση. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ και με τα χαράς ε, θα δώσω το προεδρία στην κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Ζητά συγγνώμη Πρόεδρος για τον τρόπο με τον οποίο προφέρει το όνομά σας. Παρακαλώ κυρία Παπαδοπούλου. She's going to be the moderator to... Η οποία θα είναι η συντονίστρια στο επόμενο πάνελ. Ε, ευχαριστώ όλους. Καλησπέρα σε όλους. Όπως θα ακούσετε, λέγομαι Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Κατάγομαι από την Κύπρο. Η προφορά των ονομάτων είναι πάντα δύσκολη, επομένως ζητώ συγγνώμη και εγώ εκ των προτέρων εάν κάνω κάποια λάθη με την προφορά των ονομάτων των ομιλητών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ματσόνη και τον κύριο Γκέμεση για την εισαγωγή που έκαναν σε αυτό το δεύτερο πάνελ. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα από τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, το δικαίωμα της ε, ε, ενεργού συμμετοχής στον πολιτικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι επειδή δεν υπάρχει αρκετός χώρος εδώ στο Προεδρείο, κάποιοι ομιλητές ε, θα λάβουν το λόγο από την πρώτη σειρά των εδράνων. Τους βλέπω όλους καθισμένους εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω μια εισαγωγή στο θέμα με μια σύντομη παρέμβαση των έξι περίπου λεπτών. Καλησπέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι. Ε, αυτή η ακρόαση που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ευκαιρία στις αρχές του 2013 Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών να μπορέσουμε να ε, συγκεράσουμε πολιτικές, εμπειρογνώμονες και την κοινωνία των πολιτών για να συζητήσουμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια να γίνει απτή πραγματικότητα στη ζωή των πολιτών σε καιρούς οικονομικής, ε, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης και μόνο ένα χρόνο πριν από τις επόμενες ευρωεκλογέ, ε, ο διάλογος αυτός αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου η ευρωπαϊκή ηθαγένεια να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής μας ατζέντα. Είναι ένα πολύ απαραίτητο βήμα προς μια βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με ισχυρή δημοκρατική νομιμότητα. Αυτό είναι ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών ε, για το 2013 και εγώ είμαι συγγήτρια για την έκθεση αυτή εξ ονόματο τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αλήθεια ότι η συνέχεια τη έκθεση ε, για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια του 2010 και τα αποτελέσματα τη δημόσια διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια αποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο σε αρκετού τομεί, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προσκόμματα και χρειάζονται δράσει προκειμένου να άρουμε αυτά τα προσκόμματα, ώστε οι πολίτε να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρω τα ευρωπαϊκά του δικαιώματα. Είναι λοιπόν ικανή και να εισακούσουμε τους πολίτες, να τους ζητήσουμε να μας μιλήσουμε, να βοηθήσουμε την ενεργό του συμμετοχή στον πολιτικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εφαρμόσουμε ε, διάλογο μεταξύ των πολιτών και να υπάρχει μια αυθεντική πολιτική ε, σφαίρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν οι πολίτες να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η δεύτερη σημαντική ημερομηνία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών η συνθήκη της Λισαβόνας ζητά από τους πολίτες να δημιουργήσουν διάλογο με τη θεσμικά όργανα, ζητά από τα θεσμικά όργανα συγγνώμη, να δημιουργήσουν διάλογο με τις πολίτες. Ο διάλογος θα πρέπει να αποτελεί καθημερινή αρχή και να αποτελεί και τη βάση οποιασδήποτε απόφαση λαμβάνεται. Οι πολίτες θα πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα όλες τις αποφάσεις που γίνονται εκ μέρου τους και πρέπει να πληρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και αυτών που χαράσουν πολιτική στις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες και ε, ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής οι οποίες να μεταδίδονται στο διαδίκτυο για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό ε, θεμελιώνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη συμμετοχική δημοκρατία και θα βοηθήσει να βρεθούν λύσεις στις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών και θα βοηθήσει τα δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής τους στις επόμενες ευρωεκλογές του 2014. Το δεύτερο πάνελ θα επικεντρωθεί στη συμμετοχική δημοκρατία και στα πολιτικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Το επίπεδο ε, ενεργού συμμετοχής των πολιτών αποτελεί ένδειξη του πόσο υγιής είναι η δημοκρατική ολοκλήρωση, πόσο καλά λειτουργεί η δημοκρατία και πώς η κοινωνική συνοχή ε, οικοδομείται ε, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές η συμμετοχή ήταν πρόκληση. Στα περισσότερα κράτη-μέλη λιγότερο από το 50% των πολιτών προσέφηγαν στις κάλπες και λιγότερο από το 20% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι μπορούν να επηρεάσουν προσωπικά την ευρωπαϊκή διαδικασία. Το δικαίωμα ψήφου και ε, το δικαίωμα να είναι κάποιο υποψήφιο στι τοπικέ και δημοτικέ εκλογέ είναι τρόπο ενεργού συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι και ένα τρόπο να νιώθει κάποιο ότι αφομοιώνεται στην κοινωνία, στη χώρα ε, διαμονή του. Ε, στη διάρκεια αυτού του δεύτερου πάνελ λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι καταρχάς να συζητήσουμε τη σημασία της ενεργού συμμετοχή των πολιτών ε, στον δημοκρατικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την ενθαρρύνουμε και δεύτερον να βρούμε τρόπους για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία. Τρίτον, να ενισχύσουμε τη λογοδοσία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και επιπλέον θα επικεντρωθούμε και στην, στη στέρηση του δικαιώματος ε, ψήφου ε, στις εθνικές εκλογές για όσους διαμένουν σε άλλη χώρα ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα και ε, θα συζητήσουμε τι προσκόμματα αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι πολίτες και δεν μπορούν να παλάβουν του δικαιώματος ψήφου. Ε, στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης το 62% όσων απάντησαν δήλωσαν ότι δεν υπάρχει καμία αιτιαλογή για τη στέρηση αυτού του δικαιώματος και επομένως θα προσπαθήσουμε να βρούμε ε, ποιες είναι οι καταλληλότερες λύσεις προκειμένου να επιληθεί και το συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές μας θα ήθελα να προσθέσω τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών αφορά την Ευρώπη, αφορά όλους μας ως Ευρωπαίους. Θα πρέπει λοιπόν να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, να μιλήσουμε, να δράσουμε από κοινού, να δημιουργήσουμε συνέργειες, να συμμετέχουμε και να διαβιβάσουμε το μήνυμα ότι ανήκουμε στην ίδια οικογένεια και αξίζουμε το δικαίωμα να απολαμβάνουμε την ευρωπαϊκή μας ηθαγένεια παντού χωρίς καμία διάκριση. Ελπίζω λοιπόν αυτό το δεύτερο πάνελ και όλες οι ανοιχτές συζητήσεις ε, που θα γίνουν στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών να ενισχύσει το κοινό μας όρομα για μια καλύτερη και βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με ισχυρή δημοκρατική στήριξη. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών να ε, χαράξει μια νέα εποχή για τη συμμετοχή των πολιτών στο δημοκρατικό βίο και τις δημόσιες υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβλέπω σε μια καρποφόρα συζήτηση. Ο πρώτος ομιλητές ε, είναι ο Αντώνιο Λόπεθ Ρις Βουάιτ. Νομίζω όμως ότι θα αργήσει λίγο, γι' αυτό θα δώσουμε τώρα το λόγο στο γύρο Γιώνεκ Πόλετ, ο οποίος είναι αναπληρωτής γενικός γραμματέας του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Κύριε Πόλεκ, έχετε το λόγο, Πόλετ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους Ουρανωτές αυτής της κοινή ε, συνεδρίασης η οποία αφιερώνεται στη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σημαντικό θέμα και σε πέντε λεπτά θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι κάνουν οι σοσιαλιστές πάνω σε αυτό το θέμα σε μια δύσκολη περίοδο τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ένα χρόνο μάλιστα πριν από τις ευρωεκλογέ. Σημαντικές για όλους όσοι είναι εδώ στο βήμα και για όλους εσάς φαντάζομαι και ε, δυσκολεύομαστε, δυσκολεύομαστε να κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη και γενικά οι εκλογές κίνονται σε ένα κλίμα γενικά διαφορές. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις πρέπει να αναλάβουν αυτό το έργο και είναι σημαντικό αυτό το διακύβημα για το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης. Τώρα, θα κάνω μια περίληψη έτσι γρήγορα. Ε, ένα, έχουμε πολιτικοποίηση της ευρωπαϊκής σκηνής και φυσικά να ενισχύσουμε και τη συμμετοχή. Τώρα, για την πολιτικοποίηση που είμαστε στην πολιτική ζωή, μας φαίνεται απλό. Είναι δεδομένο. Τον... Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά αυτό για έναν πολίτη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Για αυτούς στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι λίγο πολύ όλοι είναι το ίδιο. Ενώ τώρα βρισκόμαστε σε μια πολιτική κατάσταση όπου υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά και αυτό πρέπει να το δείξουμε έχουμε να κάνουμε σε ένα κλίμα το οποίο σχετίζεται με την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και βλέπουμε ε, τα πολιτικά κόμματα έχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εμείς σαν σοσιαλιστές έχουμε μια προσέγγιση η οποία στηρίζεται αυτό να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη, να βγούμε από μια πολιτική λιτότητα, να προτείνουμε, συγγνώμη, λύσεις και να προωθήσουμε την ανάπτυξη, μάλλον την απασχόληση στους νέους πραγματικά παίρνει διαστάσεις φοβερές, τρομερές σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το πρόβλημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε να έχουμε εναλλακτικέ λύσει. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο, η προσωποποίηση θα λέγαμε. Για πολλού πολίτε δεν καταλαβαίνουν ποιο εκπροσωπεί τι ο ΑΒ, τι γίνεται ακριβώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2014 θα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή διότι κάθε πολιτική ομάδα Ευρωπαϊκή θα παρουσιάσει ένα υποψήφιο για την Προεδρία της Ευρώπης. Ε, εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα κοινό υποψήφιο για τις εκλογές της Ευρωπαϊκής και αυτό είναι υπέρ, είναι σημαντικό για τις εκλογές. Θα έχουμε έναν ή μία υποψήφιο, είναι μια διαδικασία για τον ορισμό. Αυτή η διαδικασία είναι δημοκρατική και ανοιχτή. Θα αρχίσουμε το φθινόπωρο και μάλλον Γενάρη-Φλεβάρη θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Θα συμμετάσχουμε λοιπόν σε αυτή τις εκλογές ε, και με ένα κοινό υποψήφιο. Το τρίτο θέμα τώρα είναι συμμετοχή. Είναι σημαντικό να κινητοποιήσουμε τους πολίτες. Εμείς σαν σοσιαλιστές έχουμε προσπαθήσει να ξεκινήσουμε κάποιες πρωτοβουλίες, μια εκστρατεία, ε, ε, μια καμπάνια που έχει να κάνει με την φορολόγηση της διακίνησης των κεφαλαίων Επίσης τα θέματα που έχουν να κάνει με την νεολαία. Κάποιες εγγύσεις εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο, για το οποίο έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια και γίνεται μια διαδικασία και στα πλαίσια του Συμβουλίου. Αυτά είναι τα προσφυλή μας θέματα. Δυστυχώς σε πολλές χώρες υπάρχει τάση μια μειωμένη συμμετοχή. Το έχουμε δει αυτό. δίνει κανείς τη δυνατότητα συμμετοχής στις τοπικές εκλογές, αλλά στις ευρωεκλογές είναι πολύ μειωμένη η συμμετοχή. Και θα κλείσω, τηρώντας τα πέντε λεπτά, λέγοντας σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό στις πολιτικές ομάδες να δείξουν τις διακρίσεις που έχουμε ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά. Διότι στη συγκυρία που περνάμε είναι επίγον γιατί βλέπουμε ε, οι παλιοί ευρωπαϊκοί δαίμονες να ξυπνούν. Ο λαϊκισμός, Φερρυπίν, μεγαλώνει και κερδίζουν όλο και πιο μεγαλύτερα ποσοστά. Είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στο πολιτικό χάρτη της Ευρώπης. Οι εθνικισμοί που παίρνουν όλο και μεγαλύτερη διάσταση. Εμείς είμαστε λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι δημοκράτες, εμείς η οι οποίοι πρέπει να δώσουμε εναλλακτικέ λύσεις, ούτω ώστε ο Ευρωπαίο πολίτη να έχει επιλογέ και να κάνει τι επιλογέ του εν ώψη των ε, επικείμενων ευρωεκλογών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πολέτ. Σήξατε πολλά σημαντικά θέματα, πολιτικά, νέη ανεργία, συμμετοχή, πολλές ιδέες του προγράμματος δράσης και θα μπορέσετε περαιτέρω να απαντήσετε ε, στο, στις ερωταπαντήσεις. Τώρα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αντώνιο Λόπεθ της Τούρις Γενικό Γραμματέα της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού, Λαϊκού Κόμματος, του ΕΛΚ. Ε, βεβαίως υπάρχει ισπανική μετάφραση. Θα μιλήσω ισπανικά. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επίτροπο Vivian Redding για την εξαιρετική προσπάθεια που κάνει ε, για τη διοργάνωση αυτών των ημερών. Είναι θεμελιώδη σημασίας ε, τα όσα γίνονται ε, για την Ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είναι εδώ παρέντες για να μιλήσουν για το θέμα της πολιτικής συμμετοχής ε, στις επόμενες εκλογές ε, με ορίζοντα τις επόμενες ευρωεκλογές του 2014 που όπως είπε και ο συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα μια πολύ σημαντική στιγμή ως ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας πραγματικής δοκιμής. Ε, θα φανεί εάν στις επόμενες ευρωεκλογές θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την πραγματική πολιτική εκπροσώπηση των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό ε, σημαίνει ότι οι ευρωεκλογέ θα πρέπει να σταματήσουν να είναι ε, οι εκλογές ε, στις οποίες ε, το θέμα συζήτησης θα είναι απλώς και μόνο εθνικό. Εγώ ως Ευρωβουλευτής είμαι βέβαιος ότι το 80% της συζήτησης ήταν στις προηγούμενες εκλογικές ε, για εθνικά ζητήματα. Ελπίζουμε στις επόμενες ευρωεκλογέ τουλάχιστον ένα 10-15% να αυξηθεί και να προκύψει να είναι και αυτό ευρωπαϊκή συζήτηση, κάτι το οποίο είναι θεμελό η εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν έναν ίδιο χάρτη πορείας ε, όσον αφορά τα μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης να προκύψει και μία συζήτηση σε ιδεολογική βάση μεταξύ σοσιαλιστών και ε, χριστιανοδημοκρατών και να μην είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο παράδεισος των ακραίων ριζοσπαστικών στοιχείων που προσπαθούν να ε, κατακεραυνώσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα το οποίο αγαπούμε όλοι. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ σαφή διάκριση ε, για το ποια, ο, τι είναι ο, εκρο, ε, ο εξτρεμισμός, ε, τα ακραία φαινόμενα είτε αριστερά είτε δεξιά και ο ευρωσκεπτικισμός. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι ο ευρωσκεπτικισμός εκφράζεται και με κάποιο επίπεδο κριτικής και με μια δυνατότητα να προσπαθήσει κάποιος να επιτύχει το όνειρο. Δηλαδή να είναι ο Ευρωπαίος πελίτης ένας πραγματικός ε, φορέας ε, δράσης. Και νομίζω ότι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πραγματικά εκπροσωπούμε τους πολίτες, είμαστε αυτοί οι οποίοι εκλεγόμαστε από τους Ευρωπαίους πολίτες και υπάρχει δυνατότητα απόφασης και επιρροής από πλευράς μας στα γεγονότα. Όχι μόνο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ίδιο ισχύει και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως ε, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουμε μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα, παρουσία μας ε, ε, σε όλες τις χώρες στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατεία και να στηρίξουμε τα πολιτικά κόμματα τα οποία θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα στοιχείο ενημέρωση στη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία. Εμεί θέλουμε τα κράτη-μέλη ε, να είναι τα οχήματα των ευρωπαϊκών ε, πολιτικών. Εγώ είμαι από τους υπέρμαχους της επικουρικότητας. Ε, αντί να αποφασίζω εγώ, θεωρώ ότι οι σύμβουλοι του Δήμου, οι υπουργοί, οι υπουργοί των αυτόνομων περιοχών τη χώρα μα, να είναι αυτοί οι οποίοι θα μιλούν για την Ευρώπη. Και όχι μόνο στη διάρκεια των ευρωεκλογών, αλλά και στι τοπικέ του εκλογέ και στις περιφερειακέ του εκλογέ και να μην γίνεται συζήτηση μόνο για τα ευρωπαϊκά ταμεία αλλά και για άλλα ζητήματα. Αλλά και η συζήτηση για τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν πράγματι τους Ευρωπαίους πολίτες και ελπίζω ε, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι, χριστιανοδημοκράτες να δούμε ποια θα είναι τα θέματα που θα επικεντρώσουμε την προεκλογική μας εκστρατεία, να είναι θέματα τα οποία ενδιαφέρουν πραγματικά τους Ευρωπαίους πολίτες και να μην χαθούμε σε συζητήσεις οι οποίες ε, ορισμένες φορές γίνονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν δικαιολογούν ε, ε, ε, την ύπαρξή τους, δεν αποτελούν κίνητρο ούτε ε, προσεγγίζουν τους Ευρωπαίους πελίτες. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με ευγενή άμυλα μέσα στο ιδεολογικό μας πλαίσιο, αλλά πάντα με γνώμονα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι το θεμελιώδη στοιχείο σε αυτές τις εκλογές. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, σας ευχαριστώ πολύ και το ΕΛΚ είναι στη διάθεση ε, όλων ε, και των υπολείπων και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας, ευχαριστούμε και εμείς κύριε Λόπεζ, Ιστούρις White. Πράγματι, του χρόνου θα γίνει μεγάλη δοκιμή γιατί θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός των ψηφοφόρων που ψηφίζουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει οπωσδήποτε να προβληθούν περισσότερα τα ευρωπαϊκά θέματα. Ο συνάδελφός μου εκ δεξιών είναι ο κύριος Χάιντς Μπέκερ, Ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής Αναφορών. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος του ΕΛΚ και της Επιτροπής Αναφορών Έχω την εμπειρία της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών πολύ συγκεκριμένα. Είμαι από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους και μόνο μέσω της ιδιότητας του της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας μπορεί κάποιος από τους πολίτες αυτούς να ζητήσει τα δικαιώματά του μέσω της Επιτροπής Αναφορών και μάλιστα κατά πρόσωπο ε, προσωπικά ε, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να προβάλλουμε στη δημοσιότητα διότι ε, πρέπει να απολογίσουμε ότι δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να πλησιάσουμε πρόσωπο με πρόσωπο, δηλαδή ατομικά τους πολίτες. Και αυτό είναι το βασικό μας ε, μέλημα τα επόμενα χρόνια. Ακούσατε πολλά παράπονα, πολλά αρνητικά στοιχεία. Εγώ όμως ε, θέλω να μιλήσω περισσότερο για τις προτεραιότητες της ε, υλοποίησης, της εφαρμογής. Βεβαίως πρέπει να ασκούμε αυτοκριτική και χαίρομαι που και η Κομισιόν δεν καλύπτει, δεν ε, αγνοεί αυτής, αυτές της επικρίσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ίσα ίσα τις αναφέρει. Εγώ είμαι πεπισμένος Ευρωπαίος, είμαι πεπισμένος ε, Ευρωπαίος πολίτης, αλλά δεν το βλέπουν υπό αυτό το πρίσμα και, τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων. Νομίζουν ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι το α, το β, το γ, δεν ξέρουν ακριβώς τι εννοούμε. Όταν αυτά τα πολιτικά δικαιώματα τα, τα συζητούμε, αλλά δεν ξέρουμε τους πολίτες μας, δεν τους γνωρίζουμε ποιοι πραγματικά είναι. Δεν φτάνει το να τα καταγράφουμε όλα σε έγγραφα ε, ε, και να αυξάνουμε συνέχεια τον όγκο των εγγράφων. Πρέπει να τα μεταφράζουμε και σε πρακτική, σε πρακτικές εφαρμογές. Τρία παραδείγματα. Πώς θα κατανοήσουν και θα ενημερωθούν για το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν έχουν μεσάνυχτα για το πώς θα μεταφέρουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα από μία ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη. Και αυτό αφορά πολλούς Αυστριακούς πολίτες. Δεύτερο παράδειγμα, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Πώς θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα δικαιώματά τους για πανεπιστημιακή εκπαίδευση όταν δεν εγκρίνονται, δεν αναγνωρίζονται διπλώματα και πτυχία, όχι μόνο σε άλλες χώρες, αλλά και στην ίδια τους τη χώρα. Παραδείγματο χάρη, ένα φοιτητή ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Γκράτ δεν αναγνωρίζεται <laughs> στο Πανεπιστήμιο της Βιέννη, ιατρική σχολή πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τις δυνατότητες ε, περίθαλψης, τις δυνατότητες ιατρικών υπηρεσιών στους Ευρωπαίους πολίτες, εάν δεν έχουν ακούσει για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας και, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ε, στα εθνικά συστήματα υγείας και πιστεύουν ότι όλα πρέπει να τα πληρώνουν ιδιωτικά, από ιδιωτικούς πόρους. Αλλά υπάρχουν και εκατοντάδες άλλα παραδείγματα. Λοιπόν, τι κάνουν για όλα αυτά τα κράτη-μέλη μας. Πώς διαχειρίζονται αυτά τα θέματα. Δεν αποφεύγω τις επικρίσεις γιατί πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη σε πάρα πολλά ζητήματα δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους και δεν έχουν κάνει το καθήκον τους. Λοιπόν, όπως ήδη ελέγχθη και σε πολιτικό επίπεδο οι ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να αποτελέσει ένα σημείο κλειδί. Έρχεται στην, σε μια εποχή εξαιρετικά κατάλληλη όπου η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Πρέπει λοιπόν με την ευκαιρία αυτή της κρίσης να εξηγήσουμε ακόμα περισσότερο στους Ευρωπαίους πολίτες ε, τι ρόλο μπορεί να παίξει για το ξεπέρασμα της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει. Πρέπει να τους πούμε από μόνο του και τώρα αγαπητέ πολίτη έχει τη δυνατότητα να αποτανθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσει τα δικαιώματά σου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε, να πείσουμε τους πολίτες να ψηφίσουν όπως επίσης και στην εκλογή ε, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί νομίζουν ότι θα καθιερώσουμε ένα σύστημα προεδρικής, ε, προεδρικών εκλογών όπως ε, του, Γάλλου, του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Αλλά πρέπει να προσδώσουμε μια εντελώς αντίθετη, μια, μια εντελώς καινούρια ποιοτική και ποσοτική διάσταση όσον αφορά τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα μπορέσουμε να συγκινήσουμε, να φορτίσουμε συγκινησιακά τους Ευρωπαίους πολίτες άμα δεν τους γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν όλες οι ιδέες που έχουν τεθεί επιτάπητος ήδη δεδομένου ότι υπάρχει ήδη ένα ήπιο δικαίωμα ε, βέτο των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά θα πρέπει λοιπόν να ενημερώνονται άμεσα για τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς στα εθνικά κοινοβούλια και να υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών, των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Εδώ δεν υπάρχει καμία διασύνδεση, δεν υπάρχει καμία θεσμική ε, υποδομή για την ε, ε, επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίων σε επίπεδο επιτροπών. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω τρία πράγματα. Πρώτον, επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία. Αυτή την έκκληση κάνω στα κράτη-μέλη. Όχι να συμφωνήσουν σιωπηλώς, αλλά να ενεργοποιηθούν δραστήρια και με πράξεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέκερ. Πάρα πολύ ε, ε, θερμή συζήτηση και με πάθος λοιπόν. Επικοινωνία επιτρίας, επιτρία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Ζακλίν Κότεριλ, Βρετανή υπήκος συντάκτρια αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, η συντάκτρια ζει στην Ισπανία ε, και δεν μπορεί να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές εκλογές. Κυρία Κότρελ, έχετε 10 λεπτά. Καλησπέρα. Α, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που με κάλεσε σήμερα να μιλήσω για την αναφορά που έκανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, το, για τη στέρηση του δικαιωμάτου ψήφου. Είμαι Βρετανή και έχω ζήσει στην Ισπανία 23 χρόνια ε, εκμεταλλευόμενη του δικαίωμα ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση. Έχω λοιπόν το δικαίωμα να ζω και να εργάζομαι στην Ισπανία. Ε, και επίσης το δικαίωμα να ψηφίζω στο, στις δημοτικές ε, εκλογές ε, και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και ζουν πάρα πολλοί Βρετανοί απόδημοι στην Ισπανία. Λοιπόν, εγώ διδάσκω αγγλικά στους τοπικούς συμβούλους και μου είπαν ότι θα πρέπει να εγγραφώ στο Δήμο, να συμπληρώσω χαρτιά, ε, για να μπορέσω να ψηφίσω σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο. Ε, όπου έχουν γίνει αυτά έχουμε δει πραγματικά να αυξάνεται η συνδυτοποίηση της ευρωπαϊκότητας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην Ισπανία. Αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο αυτό. Στην περιοχή όπου ζω η τοπική πολιτική έχει βοηθήσει την ενσωμάτωση. Δυστυχώς όμως τα τελευταία 8 χρόνια... Ε, έχασα το δικαίωμα να συμμετάσχω στις Βρετανικές εκλογές επειδή έχω λείψει από τη Βρετανία 15 χρόνια και υπάρχει αυτός ο κανόνας των 15 ε, ετών που, που ισχύει για χιλιάδες, ε, δεκάδες χιλιάδες Βρετανών αποδήμων που ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά επειδή έχουν λείπει τόσα χρόνια από την χώρα καταγωγή τους δεν μπορούν να ψηφίσουν ε, και έτσι στερούνται τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Έχουν λοιπόν γίνει ένα σωρό αναφορές για αυτό το θέμα στην Επιτροπή Αναφορά, ο Αναφορών, παράπονα στην Κομισιόν ε, και βεβαίως το θέμα αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτή η ευρωπαϊκή κίνηση πολιτών που λέγεται Let me vote, άφησέ με να ψηφίσω. Και αυτό δεν αφορά μόνο Βρετανούς, αλλά και απόδημους άλλες ή ομογενείς άλλων ε, υπηκοτήτων. Επίσης έχω τρεις κόρες οι οποίες ε, συνυπογράψει αυτή την αναφορά και αυτές, ε, τα παιδιά μου αυτά, πάλι λόγω του κανόνα αυτού των 15 ετών, δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να ψηφίζουν εθνικά σε καμία χώρα. Πώς είναι δυνατόν. Λοιπόν, να πείσουμε τους νέους αυτούς να πιστέψουν στην Ευρώπη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καλό στοιχείο ε, και όταν, όταν υποτίθεται ότι διδάσκουμε πολυπολιτισμικότητα, γλωσσική, υποεπικυλομορφία, ανοχή, θρησκευτική κλπ. Όλα αυτά τα ωραία δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε το δικαίωμα στους ε, ψηφοφόρους να ψηφίζουν καθολικά ε, και δεδομένου ότι η ανεργία των νέων αυτή τη στιγμή θίγει πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης ε, τα, η νεολαία, η ευρωπαϊκή νεολαία έχει μεγάλους φόβους για τη μελλοντική εξέλιξη της παιδείας, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν έχει αναγνωρίσει η Κομισιόν το 2010 στην έκθεση για, τους Ευρωπαίους, ε, για την Ευρωπαϊκή Σαγένεια. αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και έχει συζητήσει το θέμα με πολλούς ευρωβουλευτές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που ε, αντιμετωπίζουμε πάλι οι ευρωπαϊκές εκλογές δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Θα πρέπει να απαλληφθούν τα χρονικά όρια τα οποία δημιουργούν αρνητικές διακρίσεις βάσει του τόπου κατοικίας και να εδρεωθούν πραγματικά δημοκρατικά δικαιώματα για όλο το, τα άτομα τα οποία διατηρούν οικονομικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς με τις χώρες καταγωγής τους και οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν ας πούμε στις βρετανικές κοινοβουλευτικέ εκλογές. Εμείς και φοροπληρώνουμε και δουλεύουμε στην Ισπανία και είμαστε και δραστήρια μέλη της κοινότητας, πολιτικά δηλαδή δραστήρια μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές και εθνικές αποφάσεις των αρχών της Ισπανίας επηρεάζουν ε, τη ζωή μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Εγώ είμαι τοπικός ε, σύμβουλος ε, και όπως σας είπα πρέπει να σέβομαι τους νόμους της χώρας αυτής στην οποία δεν έχω το δικαίωμα να ψηφίσω εθνικά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στους απόδημους Βρετανούς να ψηφίζουν ε, στη χώρα καταγωγή τους στη Βρετανία ή σε άλλους απόδημους στη χώρα καταγωγή τους και το... Πριν ε, ταξιδέψω και έρθω σήμερα έλαβα ένα email με έναν από τους πολίτες ε, του Δήμου μου και μου είπε ότι μετά από 25 χρόνια θα πρέπει επιτέλους να έχουμε φωνή σε αυτά που μας επηρεάζουν στην καθημερινή μας ζωή και στο μέλλον μας εδώ στην Ισπανία. Και πιστεύω ότι πολλοί απόδημοι αισθάνονται το ίδιο. Αυτό ήταν το μήνυμα που έλαβα. Και βεβαίως και οι κόρες μου πιστεύουν ακριβώς ε, το ίδιο. Θα ήθελε και η, η κόρη μου που είναι ενήλικη δηλαδή να μπορεί να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, ε, δύο εθνικές ε, εκλογές που θα γίνουν στην Ισπανία. Αλλά μου λέει ότι <coughs> στερούμενοι του δικαιώματο ψήφου αισθάνομαι ότι είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Έχω δηλαδή, υφίσταμαι δηλαδή διακρίσεις. Η ελευθερία κυκλοφορία, εγκατάσταση διαμονή, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η περίθαλψη, η υγεία, η παιδεία και όλα τα κοινωνικά δικαιώματα είναι πολύ ωραία και καλά, αλλά τι ισχύ έχουν όταν δεν μπορούμε να ασχίσουμε τα βασικά δημοκρατικά μας δικαιώματα εμείς είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν θα πρέπει να απαρνηθούμε την ισπανική υπηκότητα για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Ε, απορρίπτω αυτή τη λεγόμενη λύση για να μπορούμε δηλαδή να ψηφίζουμε από την Ισπανία να μην είμαστε Ισπανοί υπήκοοι ή να έχουμε διπλή υπηκότητα. Θα πρέπει λοιπόν να επεκτείνουμε το δικαίωμα ψηφοφορία και να καλύψουμε όλους αυτούς οι οποίοι ζουν σε μια άλλη χώρα από αυτή τη καταγωγή του. αλλά να μπορούν να ψηφίζουν σε εθνικέ εκλογές τη χώρα καταγωγής. Αυτή Μία τέτοια επιλογή θα πρέπει να προσφέρει τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπου ε, οι πίκοοι, οι θαγενείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισπανία θα ε, μπορούν να ψηφίζουν στην Ισπανία, επιβεβαιώνοντας έτσι με μία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ψηφίζουν σε άλλη χώρα. Ως Ευρωπαίος, Ευρωπαία υπήκος, Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ελευθερία και κυκλοφορίας. Αλλά από την προοπτική μου ως Βρετανή, ε, ε, κατοικούσα στην Ισπανία, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τεράστιες πολιτικές προκλήσεις. Εάν θέλουμε οι πολίτες να αισθάνονται μέλη της Ένωσης να ενδιαφέρονται για τις ε, λειτουργίες της, θα πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν και για τους Ευρωπαίους εκπροσώπους. Γι' αυτό ε, θα ήθελα ε, να, ε, πιστεύω και ότι η Επιτροπή Αναφορών κάνει μια ουσιαστική εργασία προς αυτήν την κατεύθυνση διότι αφήνει τη φωνή μας να ακούγεται. Ελπίζω και επίσης μπορεί να ακουστεί τα παράπονα χιλιάδων πολιτών για αδικίες που γίνονται, όπως σας πούμε περιγράφεται στην αναφορά μου. Ελπίζω ότι το έτος αυτό του Ευρωπαίου πολίτη, των Ευρωπαίων πολιτών, θα δώσει μια νέα όθηση και μέσω αυτών των ακροάσεων θα μπορέσουμε να επιτύχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Το η Ευρωπαϊκή Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν δείξει ότι ακούνε και έχουν αναγνωρίσει τις πολλές φωνές αυτές που ακούγονται για την ε, αναθεώρηση της εκλογικής διαδικασίας και για την απάλληψη αυτών των εμποδίων που στερούν τα δικαιώματα στους αποδήμους να ψηφίζουν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοντερίλ. Πράγματι, είναι τραγικό και ηρωνικό ταυτόχρονα να ε, ζητούμε από τη μία στους πολίτες να πάνε να εγγραφούν για να ψηφίσουν και να σας στερείτε αυτό το δικαίωμα να ψηφίσετε στη χώρα σας γιατί διαμένετε στην Ισπανία. Θα ακούσουμε τα σχόλια και των υπολείπων ομιλητών αργότερα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την τόσο ζωντανή παρουσίαση. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Κατρίν Κεσετζιάν αναπληρώτρια διευθύντρια του Collège Européen de Paris. Διδάσκει Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκαιο και Διεθνή Επίλυση Διαφορών στο Πανεπιστήμιο ε, Παρίσι 2, στο οποίο είναι διευθύντρια ενός προγράμματος μάστερ για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Κυρία Κεσετζιάν, έχετε 10 λεπτά για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ευχαρίστη συμμετέχω εδώ μαζί σας σήμερα το μεσημέρι και θα ήθελα να σας δώσω κυρίως δύο πληροφορίες. Euh, ε, είχαν γίνει τα στοιχεία που σας δίνουν έχουν να κάνουν μια έρευνα που δεν έχουν αξία. Η έρευνα δεν έχει στατιστική αξία, αλλά έχει γίνει και ήθελα να σας ενημερώσω για αυτήν εδώ την ακρόαση. Οι φοιτητές μου είπαν ότι αν ήθελε πραγματικά να δώσει κανείς σώμα στην ευρωπαϊκή ηθαγένεια και οι περισσότεροι από αυτούς είναι ε, Ευρωπαίοι πολίτες και είναι ειδικοί θα λέγαμε στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Λέγαν λοιπόν ότι θα πρέπει να απλοποιηθούν τα πράγματα, εκπαιδευτεί ο κόσμος στη γαλλικά λέμε ότι δεν είναι τόσο η επικοινωνία γιατί έχει αποκτήσει στα γαλλικά μια έτσι χρειά αρνητική αυτή η λέξη, ότι είναι περισσότερο μπλα μπλα. Δηλαδή ενημέρωση, κατάρτιση και κάτι το συγκεκριμένο. Θα σας πω φέρει τώρα μια ιστερία. Εγώ ήμουνα σε ένα αφιθέατρο, δίδασκα την εποχή που γινόταν πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και είπα στην αρχή της χρονιάς στους, ε, φοιτές μου ότι είναι στο πρόγραμμα, δεν είχε εγκριθεί ακόμα, υπήρχε το προσχέδιο και τους είχα πει κάνετε ό,τι θέλετε, εξασφαλίστε το κείμενο και είναι στο πρόγραμμά μας. Και έφτασα την πρώτη μέρα με το κείμενο που είχα 300 σελίδες από το site ε, Europe και μετά είχα το κείμενο στα γαλλικά, το συνολικό κείμενο, συν κάποια σχόλια και μάλιστα και ε, τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος που πρότεινε να ψηφίσει κανείς κατά. Και σας είχα πει, κοιτάξτε, έχετε αυτά ε, τα στοιχεία, ε, πάρτε αυτά τα στοιχεία, κόστησαν 2 ευρώ και σκεφτείτε πάνω σε αυτό το θέμα κατέληξα ε, με το κείμενο και το αποτέλεσμα της εργασίας του Κομμουνιστικού Κόμματος και μάση αυτό δούλεψα. Όταν λοιπόν είχαμε το κείμενο για το, την πληροφορία για το ψηφ, δημοψήφισμα, διαπίστωσα ότι μόνο μια εβδομάδα πριν είχε κανείς το, ο κόσμος, το ευρύ κοινό, τη δυνατότητα να αποφασίσει να πάρει θέση σε ένα τόσο αποφασιστική σημασία θέμα μια εβδομάδα πριν. Είναι δυνατό. Δεν μπορεί κανεί να διαβάσει ένα τόσο περίπλοκο και δύσκολο κείμενο. Εγώ πέρασα ένα χρόνο με τις φοιτές μου μελετώντας το και με τα διάφορα σχόλια. Καταλαβαίνετε ότι σε μια εβδομάδα δεν θα μπορούσε κανεί να πάρει θέση. Αυτό σας το έδωσα σαν ένα παράδειγμα. Λοιπόν, το δεύτερο όμως στοιχείο ε, έχει να κάνει μια πρόταση που μπορεί να σας φαίνεται λίγο μπανάλ, αλλά είναι ουσιαστικά η απάντηση σε αυτά που ακούμε σήμερα από το πρωί και σε σχέση με αυτά που μου είπαν οι φοιτητέ μου. Η πρόταση αυτή είναι η εξή. Στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμέσως μόλις ένας πολίτης ενοικιώνεται να του δίνει κανείς ένα εκλογικό βιβλιάριο ευρωπαϊκό. Και το σκέφτηκα αυτό από τη στιγμή που είδα αυτό το, που το κρατώ στα χέρια μου βλέπετε, το οποίο το πήρατε όλοι σήμερα το πρωί. Αλλά ε, οι ψηφοφόροι μας, οι Ευρωπαίοι όταν ψηφίζουν δεν έχουν καμιά ενημέρωση. Κοιτάξτε το αυτό εδώ. Ίσως κάτι τέτοιο να ήταν μια καλή πρόταση με συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι σημαίνουν οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι κρίμα. Διότι μειώνεται συνεχώς σε, στις Χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο για να αλλάξει αυτή η τάση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι. Σε αυτό το θα έλεγαμε εκλογικό, ευρωπαϊκό εκλογικό βιβλιάριο τι θα πρέπει να έχουμε. Σίγουρα. Δεν χρειάζεται κιόλας να να είναι και σαν χαρτιά. Μπορεί κανείς να έχει ένα στικάκι φέρπλη. Με πληροφορίες οι οποίες άμεσα μπορούν να είναι ε, χρησιμοποιήσιμες για τα δικαιώματα του πολίτη. Ειλικρινά, εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου ενημερωμένη, θεωρώ ότι το να μιλήσει κανείς ε, με σαφήνεια τι ακριβώς γίνεται στην Ευρώπη, ποια είναι τα κόμματα, τα πολιτικά, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα εθνικά και τα ευρωπαϊκά κόμματα, πραγματικά είναι δύσκολο. Ε, ε, ειλικρινά, ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση. Ξέρει ίσως για τα πολιτικά κόμματα σε εθνικό επίπεδο, αλλά τι ακριβώς γίνεται σε ευρωπαϊκό, κάπως εκεί υπάρχει μια άγνοια δεν βλέπει το σχετισμό ανάμεσα στα εθνικά και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Επίσης θα πρέπει και αυτό οπωσδήποτε να δοθεί ε, περισσότερη ενημέρωση για την ισχύ, την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, από την αρχή, όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε ουσιαστικά καμία εξουσία και από αυτό υποφέρει θα λέγαμε. Αυτή είναι η ιστορία του. Και, και πραγματικά πολλοί κόσμος δεν πιστεύει ότι έχει κάποια ιδιαίτερη εξουσία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μην μιλάει ίσως κανείς αφηρημένα, να προσπαθήσει να εξηγήσει ε, συγκεκριμένα. Να το κάνει απτό. Δεν ξέρω ο κόσμος τι ψηφίζονται νόμικοι. Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένα τρίτο στοιχείο τώρα είναι σε αυτό το βιβλιάριο θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες ε, να που έχουν να κάνουν ε, ε, ε, παραδείγματα συγκρίσιμα, να δει κανείς πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, πώς ακριβώς λειτουργεί η ψηφοφορία. Ότι υπάρχουν ε, ε προεκλογικές εκστρατείες, η διάρκεια τους, τρεις-τέσσερις σελίδες για αυτά, για να μπορεί να καταλάβει κανείς πώς ακριβώς γίνονται ευρωπλογές σε κάθε χώρα. Ε, σας το λέω αυτό, είναι μια απλή πρόταση. Εγώ επαναλαμβάνω είμαι ενημερωμένη, αλλά παρόλα αυτά το πώς ακριβώς γίνεται σε κάθε χώρα, πραγματικά δεν θα ήμουν σε θέση να σας το εξηγήσω. Τώρα τρίτη, τέταρτη πληροφορία, δεν ξέρω πού είμαι στη σειρά, στην απαρίθμηση. Αυτό που θα σας έλεγα, το στιχάκι ενδεχομένως, ο νέος, η νέα που θα πάει να ψηφίσει θα μπορούσε να ε, έχει την πληροφορία ε, της χώρου διαμονής και, και εκεί να, αμέσως να εμφανίζονται ε, σε ποιον, οι πληροφορίες που ακριβώς πρέπει να πενθυθεί κανείς σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια μεσότητα δηλαδή στην ενημέρωση αμέσως δηλαδή το άτομο να, βρει το σημείο αναφοράς. Και τελευταία πληροφορία. Ε, ειλικρινά αυτές είναι τώρα μια, οι πρώτες ιδέες που σας λέω. Τελευταία λοιπόν πληροφορία θα πρέπει όντως να εξηγεί κανείς στην πράξη τι είναι το δικαίωμα ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης να αναφερθούν και τι υποχρεώσεις να σταματήσουμε με αυτήν εδώ την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά ένα χώρι, ε, χώρος, ένα ε, εμπορικό κέντρο, ένα μόλ όπου μπαίνει κανείς, έχει δικαιώματα αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει και η ευθύνη του καθενός. Αυτή η ένωση που είναι η ένωσή μας, έτσι ίσως θα μπορέσει να λειτουργήσει ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Thank you very much. If I can just simplify what you... Ευχαριστώ. Εσείς είπατε απλούστευση, ενημερώστε, εκπαιδεύστε για τα δικαιώματα, για τη... το δικαίωμα του εκλέγην και το εκλέγεστε. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ κυρία Κεσεντζιάν και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή μας, στον κύριο Ρωμάνο Σουμπιώτο, ο οποίος είναι δικηγόρος ε, στην Αγγλία, στην Ουαλία και ε, ε, επίσης το βασιλικό σύμβουλος του Βασιλικού Συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου και επίσης ειδικεύεται σε αυτό το που λέμε στέρηση δικαιώματος ψήφου. Ευχαριστώ πολύ. Την τελευταία φορά που μίλησα για το ζήτημα αυτό, ε, μίλουσα για έξι ώρες στους δικαστές του Ευρωπαϊκού Εφετείου που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοούσα και αποφάσισαν ε, να μας καταδικάσουν. Ε, εγώ εκπροσωπώ δωρεάν έναν ε, Βρετανό υπήκο, ο οποίος διαμένει στην Ισπανία και έχει χάσει το δικαίωμα ψήφου του, διότι διαμένει εκτός ε, Ηνωμένου Βασιλείου για πάνω από 15 χρόνια. Κάθε πολίτης ο οποίος φεύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο και πάει στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, να, να δουλέψει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ε, εγώ για μια νομική εταιρεία, χάνει το δικαίωμά του ψήφου. Και αυτό φυσικά παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το εκπληκτικό είναι ότι πέραν του γεγονότος της στέρυψης ε, δικαιώματος ψήφου αυτομάτως, ε, Βρετανοί πολίτες που εργάζονται στις Βρυξέλλες, στη μόνιμη αντιπροσωπεία, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν τους επηρεάζει αυτός ο κανόνας και όσοι εργάζονται επίσης στο Βρετανικό Συμβούλιο, ούτε αυτοί ούτε οι σύζυγοί τους ε, χάνουν αυτό το δικαίωμα. Αυτό είναι η Υπάρχει βέβαια κάτι επιστημονικό ε, για την επιλογή των 15 ετών. Βεβαίως και όχι. Αν δείτε τις, ε, τα πρακτικά του Κοινοβουλίου, ε, είναι αυθαίρετη η επιλογή του χρονικού αυτού Γιατί επιλέχθηκαν αυτά τα 15 χρόνια δεν γνωρίζει κανείς. Και είναι σχιζοφρενική η ιστορία αυτής της συγκεκριμένη νομοθετική πράξη. Το 1985 κάποιο έχασε το δικαίωμα ψήφου αυτομάτω. Κάποια στιγμή κάποιο είπε ότι αυτομάτω είναι λίγο σκληρό, α το κάνουμε 5 χρόνια. Και μετά ε, κάποια στιγμή ήρθε μια νέα κυβέρνηση και είπε ας το κάνουμε 20 χρόνια. Εντάξει 20 χρόνια. Μετά ξαναπήραν τα ενία οι συντηρητικοί και είπανε 15 χρόνια. Τώρα λοιπόν φτάσαμε στα 15 χρόνια χωρίς καμία επιστημονική βάση. Όταν ήρθε να με δει ο κύριο Πρέστον, λοιπόν, είπα ότι αυτή είναι κατάφορη ε, παραβίαση των ανθρωπίνων σα δικαιωμάτων, έτσι δεν είναι. Εξέτασα λοιπόν την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με εξέπληξε το γεγονό ότι από το 1976 σε μία υπόθεση Χ κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είπε ότι είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αποστερούνται οι πολίτε του δικαιώματο ψήφου του στι εθνικέ εκλογέ εάν δεν διαμένουν στη χώρα του πλέον παρά το γεγονός ότι ε, μπορεί να έχουν δεσμούς με την ε, χώρα τους, ε, δεσμούς που μπορεί να είναι η οικογένειά τους ολόκληρη, οι κατοικίες τους, μπορεί να είναι Βρυξέλλες για την εβδομάδα και να επιστρέφουν στον Ηνωμένο Βασίλειο με το Eurostar κάθε Σαββατοκύριακο. Μπορεί να αγοράζουν Βρετανική εφημερίδα κάθε μέρα και να παρακολουθούν τα νέα στη Βρετανία κάθε μέρα. Παρόλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι χάνουν το δικαίωμα ψήφου τους. Αλλά αυτό δεν είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλό θα ήταν το δικαστήριο στο Στρασβούργο να ε, είχε κάποια λογική τουλάχιστον για τα δικαιώματα ψήφου. Ποια θα μπορούσε λοιπόν να είναι η επόμενη γραμμή επίθεσης. Ως ε, ε, γνωρίζουν όλοι οι φοιτητέ ευρωπαϊκού δικαίου και πολλοί άλλοι, υπάρχει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί χωρίς να τιμωρείται επειδή κυκλοφορεί. Και ποια είναι η τιμωρία σε αυτή την περίπτωση ότι στερείται κάποιο το δικαίωμα ψήφι του. Δεν είναι τιμωρία αυτό. Οι Βρετανοί δικαστέ δεν νομίζουν, ε, δεν έχουν αυτή την άποψη. Λένε ότι το δικαίωμα ψήφου δεν είναι και τόσο σημαντικό. Όταν να το χάσει κάποιο ε, δεν επηρεάζει πια και το δικαίωμα ελευθερία κυκλοφορία. Αλλά παραγνωρίζουν την πιο βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή ότι οποιαδήποτε απαγόρευση ελεύθερη κυκλοφορία είναι απαγόρευση ακόμα και αν είναι de Δεν υπάρχει κανένα, καμία εξαίρεση για de minimis. Οποιαδήποτε τιμωρία, οποιαδήποτε κύρωση, όποια συνέπεια και αν έχει, είναι στέρηση ελεύθερης ε, κυκλοφορίας. Η, το άρθρο 45 αναφέρεται στους εργαζομένους για την ελεύθερη κυκλοφορία. Το άρθρο 49 και τα άρθρα 20-21 από τη Συνθήκη της Λισαβόνας ε, καθορίζουν την ελευθερία κυκλοφορίας. Το επιχείρημα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια ακύρωση, δεν υπάρχει εξαίρεση δε μήνυμης και τι γίνεται ε, από εκεί και πέρα. Η κυβέρνηση έχει το βάρος της απόδειξης της ε, ποινή. Τι πρέπει να αποδείξει, πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει ένας ένομος στόχος και ότι το εθνικό μέτρο είναι ανάλογο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό είναι ο πιο λογικός τρόπος για την επίτευξη του στόχου μας. Αν εξετάσουμε λοιπόν ποιος είναι ο ένομος στόχος, ε, είναι ότι αν ζούμε σε μία ένωση η οποία έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία μιας ολαιόνα και στενότερης ένωσης μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η τιμωρία, οι ποινές προς τους Ευρωπαίους πολίτες, διότι μετακινούνται ελεύθερα και χάνουν τη στέρηση του δικαιώματος ψήφους, είναι σκανδαλώδης. Είναι σκανδαλώδης. Κανείς όμως, κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό στις ε, εφημερίδες, καμία βρετανική εφημερίδα δεν αναφέρει το γεγονός. Είναι όμως σκανδαλώδες. Και επίσης, Έστω ότι υπάρχει ένομο στόχο. Και τι λέει η Βρετανική κυβέρνηση, ότι αν ε, κυκλοφορείτε εκτό Ηνωμένου Βασιλείου, χάνετε τη σχέση σα με τα βρετανικά ζητήματα και χρησιμοποιεί την λογική του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1976. Το δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, το 1976 είπε ότι δεν μπορεί να βρει κανείς εφημερίδες, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα τεκτενόμενα στη χώρα του, ε, η επικοινωνία δεν είναι και τόσο καλή, δεν ε, σας επηρεάζει άμεσα το τι συμβαίνει στη χώρα και ούτω καθεξής. Για όλα όμως αυτά τα επιχειρήματα υπάρχει μια απάντηση. Έστω ότι χάσαμε ε, το, στο θέμα του ένομου στόχου. Τι γίνεται με την αναλογικότητα. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι μόνο οι Βρετανοί πολίτες που έχουν κάποια σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να ψηφίσουν και θα πρέπει να παραμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει να χάνουν το δικαίωμα ψήφου τους ε, μόλις αποχωρήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι μόνο αυτοί που έχουν κάποια σχέση με τη χώρα ψηφίζουν γιατί να μην λέμε από τους Βρετανούς πολίτες που διαμένουν στις Βρυξέλλες να εγγραφούν στη μόνιμη αντιπροσωπεία ή στην Βρετανική πρεσβεία αν θέλουν να ψηφίσουν. Αυτό το οποίο χρησιμοποιήσω ως επιχείρημα στο δικαστήριο είναι το δικαίωμα ψήφου. Δεν είναι παθητικό δικαίωμα όπως το να λάβει κάποιος με επιταγή στο ταχυδρομείο. Είναι ενεργό δικαίωμα πρέπει κάποιο να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει να εγγραφεί για να ψηφίσει. Και όλοι γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να είναι και μεγάλο μπελά. Αλλά αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Και όχι μόνο να εγγράφονται στα Μητρώα ε, στου εκλογικού καταλόγου, αλλά από εκεί και πέρα να έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Δεν είναι παθητικό δικαίωμα, είναι ενεργό δικαίωμα. Αυτό από μόνο του συνιστά φίλτρο, διότι κάνει διάκριση μεταξύ ανθρώπων που δεν θέλουν να ψηφίσουν, επομένω χάνουν και το δικαίωμα ψήφου του, αλλά ε, μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμά του, οι Βρετανοί πολίτε που επιθυμούν να ψηφίσουν. Αυτό που λέω στους δικαστές τώρα είναι ότι η Βρετανική νομοθεσία επιτυγχάνει ε, ακριβώς το αντίθετο. Αφαιρεί, στερεί το δικαίωμα ψήφου από τους ανθρώπους που θέλουν να ψηφίσουν και δεν έχει και καμία συνέπεια για αυτούς που ούτως ή άλλως δεν θέλουν να ψηφίσουν. Τα επιχειρήματα λοιπόν είναι πολύ απλά. Ο στόχος ήταν η υπόθεση αυτή τουλάχιστον να γίνει κατανοητή από τους Ευρωπαίους δικαστές ε, και ε, καλύτερα να πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο, έχουμε χάσει στο εφετείο και ζητήσαμε άδεια να προσφύγουμε στον Άριο Πάγο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, περιμένουμε την απάντηση. Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο του ε, Ηνωμένου Βασιλείου δεν μας δώσει το δικαίωμα να καταθέσουμε έφεση, τότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα τελειώσει όλη αυτή η συζήτηση σε νομικό επίπεδο για τη στέρηση δικαιώματος ψήφου των ατόμων που δεν διαμένουν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και κάτι τελευταίο, αυτό το οποίο είναι αδιανόητο είναι ότι αντιμετωπίσαμε εμπόδια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αυτό ήταν ε, ιδιαίτερα διδακτικό διότι μου έμαθε τα πάντα για τις ε, διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί κάποιος να ζητήσει ε, δικαστική αναθεώρηση μιας πράξης. Τη ζητήσαμε, μας το αρνήθηκαν, δεν μας δόθηκε καν το δικαίωμα να αναθεωρηθεί η νομοθεσία δικαστικός. Ο δικαστής στην ε, καρέκλα του, στον κήπο του τον Αύγουστο αποφάσισε ότι δεν ήταν και τίποτα σημαντικό. Κατα... Παρανόησε τελείως τα της υπόθεσης. Εμείς νόμιζα ότι λέγαμε ότι το, ε, η Ευρωπαϊκή Συνθήκη δίνει δικαίωμα σε τρίτους υπηκόους να ψηφίζουν στις κοινοβουλευτικέ εκλογές. Ενώ εμείς λέγαμε ότι στερείονται το δικαίωμα ψήφου εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι τελείως διαφορετική υπόθεση αυτή. Έγινε μια κρόαση ενώπιον ε, του κυρίου Σμίτεν, που ήταν ο καλύτερος δικαστής όλων, ο οποίος μας έδωσε άδεια για δικαστική αναθεώρηση. Έγινε η ακρόαση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Χάσαμε. Και ζητήσαμε το Ανώτατο Δικαστήριο ε, δικαίωμα έφεσης. Ε, μας αρνήθηκαν γραπτός το δικαίωμα έφεσης. Είπαμε να γίνει ακρόαση, έγινε ακρόαση, δικαίωμα πλέον να εφεσιβάλλουμε την απόφαση. Περνάμε στο φετίο, γίνεται η ακρόαση, χάνουμε και πάλι και ε, γράφουμε και ζητάμε γραπτό σε επιστολή να ε, ε, απευθυνθούμε στον Άριο Πάγο και χάσαμε και πάλι και είμαστε στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας. Ζητούμε και πάλι δικαίωμα να εφεσιβάλουμε την απόφαση. Αυτά με δύο λόγια είναι τα όσα ζούμε και με μου άρεσε ιδιαίτερη η παρουσίασή σας, διότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι η σωστή λύση, γιατί υπάρχει μια απόφαση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία συνεχίζεται και προχωράει στο διηνικές. Τα επιχειρήματα του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αυτά τα οποία θα κερδίσουν, αλλά δυστυχώς οι δικαστές θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα πολιτικό το ζήτημα. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι το ίδιο φρονεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν δηλώσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το δικαίωμα ψήφου δεν εμπίπτει στι αρμοδιότητε του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό το θέμα δεν είναι ευρωπαϊκό δίκαιο. Πραγματικά λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργατα, επειδή οι δικαστές φαίνεται να διστάζουν τόσο πολύ με το θέμα αυτό, να κάνει μια πρόταση. Είναι γελίο. Εγώ είμαι πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έχω ψηφίσει ποτέ. Ψήφισα στι ευρωεκλογέ του 1979, ε, πέντε μέρε μετά που έκλεισα τα 18 και αυτό ήτανε. Ε, ζω πάντα εκτό του Ηνωμένου Βασιλείου και είμαι προϊόν μια γενιά ε, που περιγράψατε. Είμαι μισό Γερμανό, μισό Ιταλό, γεννημένο στην Ελβετία, παντρεμένο με Ισπανίδα, ζω στι Βρυξέλλε. Καταλαβαίνετε, ένα συναφίλευμα λαών. Thank you very much, Mr. Sabioto. It seems that... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σουμπιώτο. Λίγαν περίπλοκο το θέμα αυτό και πράγματι τα ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να επιληθούν τα προβλήματα. Και η κυρία Κιάρα Άνταμο είναι η επόμενη ομιλήτρια, επικεφαλής της μονάδας, Ιθαγένεια της Ένωσης, μονάδας Ιθαγένεια τη Ένωση και ελεύθερη κυκλοφορία, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη τη Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι τελευταία μελήτη αυτού του πάνελ και είμαι σε πλεονεκτική αλλά και ε, ενδιαφέρουσα θέση δεδομένου ότι πρέπει να συγκεράσω τις παρατηρήσεις που έκαναν οι προλαλήσαντε συνάδελφοι και ε, να σας ε, παρουσιάσω βεβαίω και το ρόλο της Κομισιόν μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Όπως τόνισε και Κυρία Ματσόνη, η συνθήκη της Λισαβόνας ε, περιέγραψε, οριοθέτησε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Και σήμερα το πρωί αναφέραμε επί μακρόν την, ε, τις πρωτοβουλίες ε, για τον Ευρωπαίο πολίτη, την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής βάσει του άρθρου 10 της Συνθήκης, το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική ευρωπαϊκή ζωή κάθε πολίτη και ούτω καθεξής. Η Κομισιόν λοιπόν έχει συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση παρουσιάζοντας, συντάσσοντας και δημοσιεύοντας αυτή την έκθεση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010. Και εδώ περιγράφεται, περιγράφονται τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας στο ρόλο τους ως πολιτικοί παράγοντες. Τρία στοιχεία θέλω να τονίσω. Καταρχάς η πληροφόρηση ενημέρωση των πολιτών, αυτό ήταν το σημείο κλειδί. Δεύτερον, η υλοποίηση η εφαρμογή της συνθήκης και τρίτον, κατάλληλη νομοθεσία και ενθάρρυνση των πρωταγωνιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσουν το ρόλο τους στην αύξηση της ευρωπαϊκής συμμετοχής. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτού του hearing έχουμε παρουσιάσει καινούρια μέσα ε, τα οποία ε, θα διαγράψουν το, τη μελλοντική πορεία μας και ε, πολύ λίγη, ένα πολύ μικρό ποσοστό των πολιτών μας, ε, περίπου το 1 τρίτον, είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους. Η μεγάλη πλειοψηφία, τα 2 τρίτα, ξέρουν τα βασικά δικαιώματα. Ας πούμε, ότι έχουν το δικαίωμα, του εκλέγην και του εκλέγεστε σε τοπικό επίπεδο, ότι μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές της τοπικής αυτοδίκησης όταν διαμένουν σε, μια, σε ένα άλλο κράτος μέλος. Και από τις πρόσφατες, από τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, το δικαίωμα αυτό της τοπικής ε, ψήφου δεν έχει αυξήσει, δεν έχει συμβάλει στην αύξηση της ευρωπαϊκής συμμετοχής ε, στην ψηφοφορία. Ενώ αυτός είναι ο στόχος Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ζητήσω από την Κομισιόν πάντοτε να ενισχύει τις ε, διαδικασίες ε, ε, ενημέρωσης, την κατάρτιση σε αυτά τα ζητήματα. Και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ορίστηκε το 2013 ως έτος του Ευρωπαίου Πολίτη. Από τη σκοπιά του 2010, όταν το συζητούσαμε, ήταν μια πάρα πολύ σωστή ιδέα και βλέπουμε πόσο επίκαιρη είναι φέτος, το 2013. Διότι πολλές καλές ιδέες ακούγονται από τους πολίτες μας. Κάναμε λοιπόν πέρσι και μία σφιγμομέτρηση της κοινή γνώμης, μία δημόσια διαβούλευση. Σημειώσαμε όλα τα σχόλια και τα λάβουμε υπόψη ε, στο μέλλον. Η ακρόαση αυτή είναι μια ευκαιρία για την Κομισιόν να ακούσει τις απόψεις σας από το τοπικό επίπεδο, από τη βάση, αλλά είναι ευκαιρία και για σας να ακούσετε τους εμάς. Ε, έχω πάει σε πολλά ε, δημαρχία, σε πολλές τοπικούς φορείς, έχω μιλήσει σε αυτούς, έχω ακούσει τις απόψεις τους για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ε, και η Κομισιόν, όπως ανέφερε και ο κύριος Μπέκερ, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την υλοποίηση. Βεβαίω, είναι ένας ε, κέριο ρόλος που μπορεί να ασκήσει η Κομισιόν. Ε, όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγεστε, κάποιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα, ακόμα και αν μένει σε ένα άλλο κράτος μέλος. Έχουμε λοιπόν λοιπόν ε, ε, εφαρμόσει ισχυρά μέτρα υλοποίησης όλου αυτού του θεσμικού πλαισίου Έχουμε βοηθήσει στην, ε, τον ορισμό κριτηρίων διαμονής για να αποφασίσει ένα κράτος μέλος ποιος μπορεί να έχει θέση υποψηφιότητα και ποιος όχι. Επίσης έχουμε προσπαθήσει να πλουστέψουμε τη διαδικασία υποβολής πιστοποιητικών. Βλέπετε λοιπόν δέσμοι μέτρων που επηρεάζουν συγκεκριμένα Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε συνεργαστεί λοιπόν στενά με τις εθνικές αρχές για τα, την ενίσχυση αυτή των δικαιωμάτων ψήφου και έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο. Παρό Παρόλα αυτά έχουμε δει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προσκόμματα σε Ευρωπαίους πολίτες να είτε να ιδρύσουν ε, καινούργια κόμματα είτε να συμμετάσχουν σε καθιερωμένα πολιτικά κόμματα σε αυτή την άλλη χώρα που κατοικούν. Ε, και δεν θα πρέπει να δεχθούμε μια κατάσταση όπου σημειώνονται αρνητικές διακρίσεις κατά Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας Ευρωπαίος πολίτης να γίνει μέλος, να γραφτεί σε ένα εθνικό κόμμα, ας πούμε, όπως η υπήκοη του κράτους αυτού, επειδή δεν είναι υπήκος. Πέρσι το Συμβούλιο Βούλιο υιοθέτησε την οδηγία πλούστευσης της διαδικασίας υποβολής υποψηφιότητος στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση της συμμετοχής. Πιστεύουμε ότι 8 ε, στους 10 Ευρωπαίους πολίτες θα είχαν μεγαλύτερο κίνητο να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές αν ήταν καλύτερα ενημερωμένοι Υπάρχει όμως, όπως σημείωσαν και προλαλήσαντες, αυτή η μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης. Και γι' αυτό Χαίρομαι ιδιαίτερα που προτείνεται η υποβολή υποψηφιωτήτων και η ανακοίνωση της υποβολής υποψηφιωτήτων για τη θέση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα επιτύχουμε στην ε, περισσότερη, σε μεγαλύτερη συμμετοχική δημοκρατία αν δεν μας βοηθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτό το τόνισαν ήδη οι προηγούμενοι ομιλητές. Και ο κύριος Γκέμεση από την Ουγγαρία είπε πολύ σωστά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. πριν από 15 μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισέτησε μια γνωμοδότηση για την ε, πολιτική συμμετοχή και αυτή θα την αναλύσουμε λεπτομερώς στην υπηρεσία μου. Ο κύριος Σουμπιώτο δεν θα πρέπει να ανησυχήσει ε, λέγοντας ότι ε, εάν προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα, νεκρώσει, θα νεκρωθεί η συζήτηση. Όχι, ίσα ίσα υπάρχει τεράστια πίεση από πάρα πολλές πλευρές η συζήτηση αυτή να προβληθεί η Κομισιόν. Έχει πει επανειλημμένως ότι η οργάνωση των εθνικών εκλογών έγκυται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό είναι σωστό. Αλλά λέμε ταυτόχρονα ότι εάν πολίτες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εκλογή μια εθνική κυβέρνηση, τότε του στερείται η εκπροσώπηση στο Συμβούλιο των Υπουργών. Άρα του στερείται η συμμετοχική δημοκρατική εκπροσώπηση στα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αντιτίθεται στην ελεύθερη κυκλοφορία. Ευχαριστώ κυρία Ντάμου. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου, γι' αυτό τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκέραντ Χάφερτ, μέλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων, αναπληρωτή της Επιτροπής Αναφορών. Ήταν ένας από τους εισηγητές για την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για πάνω από τρει δεκαετίες ήταν ιδιαίτερα δραστήριο σε αρκετές με κυβερνητικές οργανώσεις που προωθούν την ε, άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Έχετε πέντε λεπτά για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και να καλωσορίσω και από πλευράς μου όλους όσους ε, συμμετέχουν σήμερα σε αυτή την ακρόαση. Επειδή κατά κάποιο τρόπο έχω τον τελευταίο λόγο, θα ήθελα να ε, κάνω μια ευρύτερη προσέγγιση. Γίνεται αυτή η ακρόαση σε μια χρονική συγκυρία όπου η Ευρώπη ε, εν μέρη ε, είναι σε αναταραχή. Οι πολίτες είναι στους δρόμους, διαδηλώνουν ε, και διαμαρτύρονται και ούτε καθεξής. Και τμήμα αυτού είναι και ε, μια έκφραση του γεγονότος ότι θεωρούν ότι δεν έχουν και πολύ μεγάλο λόγο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ξεκίνησα στα αγγλικά αλλά θα ήθελα να συνεχίσω στα γερμανικά αν μου επιτρέπετε διότι θα είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να σας πω την άποψή μου και δίνει και τη δυνατότητα ξέρει τους διερμηνείς μας, λέει ο μιλητής, να με μεταφράσουν. Um, den stand der... ανησυχώ πολύ για τη δημοκρατική κατάσταση στην Ευρώπη. Είμαστε, ανησυχούμε συνεχώς με θέματα εσωτερικά της Ευρώπης και δεν φροντίζουμε την εξωτερική μας εικόνα. Έχει κανείς την εντύπωση ότι οι πολίτες δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αποφάσεις που τους αφορούν, όπως θα το επιθυμούσαν. Και αυτό είναι ο λόγος της απογοήτευσης μιλάμε για το δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογές, όπως ελέγχθη εδώ. Αυτό το δικαίωμα δεν μπορούν να συμμετάσχουν και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς του Ευρωπαίου πολίτη που επιτρέπει σε κάθε ένα, κάθε μια να ασκεί αυτό το δικαίωμα. Δεύτερον, μιλώντας για το δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να συμβάλλουμε ούτως ώστε οι πολίτες να καταλάβουν ποια είναι η σχέση από τη μια η εκλογή που κάνουν και οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολίτες ορίζουν κάποιον υποψήφιο να καταλάβουν, να δείξουν εμπιστοσύνη και να μην ψηφίζουν με κλειστά τα μάτια. να μην ε, δηλαδή διαπιστώνει, ψηφίζει κάποιον τον οποίο δεν ξέρει, δεν είναι αυτός τον οποίο έχει επιλέξει, γίνονται εγκρυπτό ε, διαδικασίες. Αυτό ίσως θα επέτρεπε, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια σχέση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ηθιγένεια και τις ε, αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει ένας εισηγητής να δει για το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Έχουμε δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Μπορούμε να πούμε θα πρέπει να γίνουν δεκτά πολιτικά κόμματα, τα οποία ήδη, μόνο τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό όμως θα οδηγούσε στην αποκλεισμό άλλων νέων κομμάτων, το οποίο όμως αποτελεί δικαίωμα του ψηφοφόρου. Γι' αυτό θα πρέπει από τη μια να αποφύγουμε να βάλουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Στην Επιτροπή μας αποσχολεί αυτό, όσον αφορά δηλαδή τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ε, έχουν ένα καθεστώς το οποίο ε, θα πρέπει να εξασφαλίζει κάποιες δημοκρατικές αρχές. Για παράδειγμα, ο Α ή Β θέλει κάποιος ε, να στείλει κάποιον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτός θα πρέπει να είναι υποψήφιος ο οποίος θα οριστεί σαν υποψήφιος από, το πολιτικό, από ένα α ή β πολιτικό κόμμα. Θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να εμβαθύνει κανείς τη δημοκρατική διαδικασία. Και όταν μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκή θαγένεια έχουμε προσπαθήσει να μειώσουμε τα εμπόδια. Θυμάστε που το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε φέρει πιέν ένα ελάχιστο αριθμό ε, πολιτών και εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να μειωθεί αυτός ο αριθμός για να μπορέσει να γίνει μια πρωτοβουλία πολιτών. Δεν είναι όμως τα πράγματα τόσο εύκολα. Δίδαμε δηλαδή ότι τη συλλογή υπογραφών ηλεκτρονικά σε μεγαλύτερο διάστημα δεν μπορούν να καλά. Οι πρωτοβουλίες των πολιτών είναι μια δύσκολη διαδικασία και εμείς έχουμε πετύχει κάτι όσον αφορά αυτό το θέμα για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει όμως να βελτιώσουμε το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό. Όπως θα έχει όμως η κατάσταση τώρα, ακούει κανείς, διαψώνει κανείς ότι λέγονται πολλά από τους πολίτες για θέματα δημοκρατίας για τεχνοκράτες και είναι σαφέστατο ο Ευρωπαίος πολίτης έχει κάτι να πει. θα πρέπει να μπορεί ο Ευρωπαίος πολίτης για τι επόμενε εκλογέ να προσεγγίσει, να έχει πρόσβαση σε όλα τα θέματα, θέματα που αφορούν τον προπολογισμό και δημοκρατικές μεθόδους υπήρχε μια διαδικασία στην οποία προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη και αμεσότερη συμμετοχή ούτως ώστε να μπορέσουμε σταδιακά να δώσουμε τη δυνατότητα στον Ευρωπαϊκό πολίτη να έχει ο ίδιος τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χέφνερ για τη συνεισφορά σας. Ε, τώρα θα ξεκινήσουμε με τον πρώτον γύρο παρεμβάσεων από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν το λόγο θα λάβουν ε, οι συμμετέχοντες αν υπάρχει χρόνος. Θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι προκειμένου να μπορέσουν να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, ο χρόνος ομιλίας περιορίζεται στα δύο λεπτά ακριβώς. Ε, μπορείτε κάλλιστα να θέσετε ερωτήσεις, να πείτε τις απόψεις σας, να κάνετε τις προτάσεις σας. Κάποια μέλη έχουν ήδη ζητήσει το λόγο. Καταρχάς, η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Και κατόπιν, ο κύριος Αντροντάφ και ο κύριος Σκάπα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά θα μιλήσω. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε του πολίτε πώ λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ούτω καθεξής. Και η περιέργεια μου είναι εξή και το θέτω προ όλου ε, τους ομιλητές. Πώς αξιολογείτε το ρόλο των γραφείων πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα ολόκληρο δίκτυο σε διάφορε χώρε ε, γραφείων πληροφοριών και θα πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για το πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο και τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε τις επιθυμίες μας και να εξετάσουμε πώς μπορούμε να δώσουμε νέα όθηση στις δραστηριότητες τους και τι ειδικέ δραστηριότητες περιμένουμε από αυτά τα γραφεία ε, το επόμενο 1,5 χρόνο πριν από τις ευρωεκλογέ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς λειτουργούν αυτά τα γραφεία και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επηρεάσουμε περισσότερο το πώς ε, λειτουργούν. Επίσης, κάτι ακόμα. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα σε περιπτώσεις όπως ε, τη άκτα που αποδεικνύουν ότι το κοινοβούλιο μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικό από τα φυλάδια στους πολίτες. Πράγματι, έχετε δίκιο. Ε, ο κύριος Άντριου Ντάφ έχει το λόγο. Για δύο λεπτά. Κοιτάξτε. Εγώ είμαι εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα της εκλογικής μεταρρύθμισης και νομίζω ότι μου επιτρέπετε να μιλήσω λίγο περισσότερο προκειμένου να εξηγήσω λίγο καλύτερα κάποια από τα νομικά και πολιτικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε προσπαθώντας να εξυγχρονίσουμε τα θεσμικά μας όργανα. Ε, όπως αρκετοί θα γνωρίζουν, προσπαθήσαμε και εγώ προσπάθησα και η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων έκανε μία απόπειρα για τις εκλογές του 2014 να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή επικράτεια για την εκλογή 25 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εκλέγονται από ένα υπερευνητικό ψηφοδέλτιο. Η λύση αυτή θα είχε ρυθμίσει την ε, αύξηση των ε, πολιτικών ε, κομμάτων, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, τα οποία θα ήταν υποχρεωμένα να συνεργαστούν πιο ενεργά ως ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, όπως δεν κάνουν αυτή τη στιγμή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αντίθετο βέβαια σε αυτό και οι σοσιαλιστές ήταν αντίθετοι και νομίζω ότι υπάρχει εκπρόσωπός τους εδώ σήμερα, αλλά και το ΕΛΚ, ε, το οποίο εκπρόσωπος εξαφανίστηκε, ήταν αντίθετη λοιπόν στην εκλογική μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό πρώτον λοιπόν. Υπάρχει ε, πολύ μεγάλη εσωτερική αντίσταση στη μεταρρύθμιση. Δεύτερον, για το θέμα της ε, παράτασης ε, του δικαιώματος ψήφου σε πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό. Ο κύριος ε, Σουμπιώτο διαμαρτυρήθηκε για τη στέρηση δικαιώματος ψήφου. Εγώ είχα προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινήσει μια έκθεση προκειμένου να δράσει βάσει του άρθρου 25 ε, της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής ε, των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας στο άρθρο 20 σημείο 2 της Συνθήκης ώστε να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις απαντήσεις τους Προ το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε. Δηλαδή να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα στερείται του δικαιώματο ψήφου σε εθνικέ εκλογέ. Ελπίζω ότι σύντομα θα μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει αίτηση για ε, πρόσβαση στην ECHR και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλου του ECHR λέει ότι τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ε, για να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους στην νομοθετική διαδικασία. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στις ευρωπαϊκές συνθήκες, αλλά εφόσον προσχωρήσουμε στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορεί να αποφασίσει σε συλλογικές αγωγές επί του ζητήματος και θα έχει πλέον ε, το περιθώριο να το κάνει. θα αποδεσμευθεί η νομολογία τους για την ελευθερία κυκλοφορίας, θα μπορούν να έχουν και αυτό το στοιχείο επιπλέον και θα υπάρχει νέο καθήκον να εφαρμόζεται απευθείας η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, στους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχει λοιπόν μια ρανίδα ελπίδας. Αλλά το πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση θα πρέπει να εντατικοποιηθεί πριν ε, μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό το τεράστιο χάσμα στο οποίο έχουμε περιέλθει κατά λάθο νομίζω και όχι η κακή την πίστη. Ήταν βέβαια κακό το λάθος, ε, μεγάλο το σφάλμα και θα πρέπει να επανορθώσουμε για την ε, για να μπορέσει να ανθίσει η μεταεθνική δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νταφ και ο κύριος Κάπαν Σούκερ για την ερώτησή του. Δύο λεπτά. Ο κύριος Σόγκορ. Ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά όχι μόνο κατά τη διάρκεια ενός ευρωπαϊκού έτος εκλογών, κάθε χρόνο και συνέχεια. Γιατί οι πολίτες με τους οποίους μιλάμε πάντοτε αναφέρονται σε τοπικά ζητήματα. Άρα λοιπόν καλή συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά τα τοπικά ζητήματα είναι τα καυτά. Έχω λοιπόν το αίσθημα μετά από όλα αυτά που έχω ακούσει από όλου ότι τα περισσότερα προβλήματα προσπαθούν να τα σπρώξουν προς την εθνική, προς την επίλυση μέσω εθνικών οργάνων και φορέων. Εδώ έχουμε προβλήματα διακρίσεων, έχουμε προβλήματα ανθρώπων που χάνουν την ε, ηθαγένειά τους, ε, προβλήματα ανθρώπων που χάνουν τις περιουσίες τους ε, ή που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα σύμβολα που θέλουν κλπ και ακούμε συνέχεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αρμοδιότητες να δράσει σε αυτά τα προβλήματα, δεδομένου ότι δεν είμαστε μόνο οικονομική ένωση. Όπως κάναμε λοιπόν με την κοινότητα των Ρωμά, γιατί δεν εκπονούμε κανονισμούς και νομοθετικές ρυθμίσεις για τους ανισαγενείς που αυτή τη στιγμή καταταλαιπωρούνται μέσα στην Ένωση. Τα τοπικά προβλήματα είναι τα πραγματικά ευρωπαϊκά, όχι αυτά τα οποία μας έρχονται ε, ε, ουρανοκατέβατα από τα υψηλά επίπεδα, από τα ουράνια. Τα τοπικά, εδώ, στη βάση, αυτά, στις ρίζες, αυτά μας ενδιαφέρουν και μας καίνε. Γιατί παραδείγματο χάρη υπάρχουν ε, αγρότες οι οποίοι υφίστανται αρνητικές διακρίσεις. Ευχαριστώ κύριε Σόγκορ, λέει πρόεδρος. Παρακαλώ υπάρχουν άλλα μέλη. No. Ε, I have two questions which have been received by Twitter. Ε, λάβαμε και σχόλια μέσω του Twitter. Μία ερώτηση που λέει μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακάμψει τις διατάξεις του άρθρου 51 του χάρτη σε δικαιωμάτων. Άλλη ερώτηση. Θέλουμε να ξέρουμε αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρη δικαιώματα ψήφου στους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν σε άλλο κράτος. Πιστέψτε με, εγώ είμαι εισηγήτρια για το θέμα το, το σημερινό, δηλαδή του, Ευρωπαίου, του έτος του Ευρωπαϊκού Πολίτη και εγώ υπεραμείνουμε ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελεύθερης διακίνησης και διαμονής. Έχουμε τόσους πολλούς κανονισμούς όσο και εμπόδια. Εάν θέλουμε πραγματικά να εδραιώσουμε αυτά τα δικαιώματα και να δείξουμε αλληλεγγύη προς άλλους Ευρωπαίους που υποφέρουν. Ε, μην ξεχνάτε, προέρχομαι από ένα νησί όπου ο μισός ε, πληθυσμός στερείται των βασικών του δικαιωμάτων διότι έχει καταληφθεί από ξένη δύναμη. Αν θέλουμε λοιπόν και στην Κύπρο να ενισχύσουμε τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει πραγματικά να δράσουμε. Ε, δίνω λοιπόν το λόγο στους, ε, στους, στα μέλη του πάνελ εδώ πριν ε, και στην κυρία Ματσόνη αν θέλει. Έχετε το λόγο για να ολοκληρώσουμε. Πολύ σύντομα, διότι η κυρία Ματσόνη που προεδρεύει είναι εδώ είναι και η κυρία Ματσόν και μαζί με την Επίτροπο Ρέντινγκ θα δώσουν μία συνέντευξη τύπου μετά τη συνεδρίαση. Και μπορείτε να μείνετε εδώ μετά την εισήγηση της κυρίας Ρέντινγκ. Θα κοιτάξω να είμαι σύντομα να πω απλώς λυπάμαι που για ένα τέτοιο θέμα δεν, μπορούμε να, δεν να έχουμε μια, ένα ευρύ διάλογο με την αίθουσα. Σίγουρα θα υπήρχαν ενδιαφέροντες ερωτήσεις σε σχέση με το... Ε, υπάρχουν δικαιώματα που μπορεί να ξανακερδίσει ο πολίτης, υπάρχουν όμως και νέα δικαιώματα. Ένα σημαντικός διάλογο σε αυτό το θέμα. Σε όλο και περισσότερε χώρε το βλέπουμε. Υπάρχει το δικαίωμα του ψήφου του ε, πολίτη σε μια άλλη χώρα για τις εθνικές εκλογές, αλλά υπάρχει και το θέμα της ελογής ε, ε, ατόμων που ζουν ε, ε, στο εξωτερικό και εκπροσωπούν τους πολίτες σε αθηνικά κοινοβούλια. Πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα σε μια Ευρώπη όπου βλέπουμε όλο και πιο πολύ κινητικότητα για διάφορους λόγους, δηλαδή για καλούς ενδεχομένως λόγους, λόγω της οικονομικής δραστηριότητας. Έχουν δικαιώματα τόσο στις χώρες υποδοχής αλλά και στις χώρες από τις οποίες κατάγονται. Για το 2014 τώρα και η σημασία των ευρωεκλογών. Υπάρχει το θέμα της ε, μειωμένης συμμετοχής. Ανέφερα ότι διαπιστώνει κανείς με λύπη υπάρχει ε, εδώ πέρα η ευθύνη της πολιτικής τάξης η οποία πρέπει να κάνει τα αυτοκριτική για τον τρόπο τον οποίο γίνεται η εκστρατεία και να πρέπει δηλαδή να προσεγγίσει κανείς τα πραγματικά ευρωπαϊκά θύματα όταν γίνονται ευρωεκλογές και όχι εσωτερική ε, αντιπαράθεση. έχει να κάνει φυσικά με τις θέσεις των κομμάτων, τη θέση τους, ποια είναι στην εξουσία, ποια όχι. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι εκλογές είναι λίαν σημαντικές για τον πολίτη στην Ευρώπη. Είμαστε σε μια οικονομική, κοινωνική δύσκολη περίοδο. Η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί. Υπάρχουν και άλλες λύσεις που πρέπει να ε, λυθούν σε θέματα με την τα δημοσιονομικά, την οικονομία, την απασχόληση, την απασχόληση των νέων. Σίγουρα υπάρχουν διαχειριεύματα για τα οποία μπορεί κανείς να κινητοποιήσει τον Ευρωπαίο πολίτη και πραγματικά ε, να μας έχετε εμπιστοσύνη. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Η κυρία Ανταμό, πολύ σύντομα παρακαλώ. ο ρόλος των γραφείων πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. δεν έχω αντίρρηση να απαντήσει η Προεδρεύουσα, αλλά βεβαίως τα γραφεία αυτά εμπλέκονται πλήρως στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, βοηθούν στην οργάνωση τοπικών συνεδριάσεων, επισκέψεων κλπ. Τώρα, εάν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεπεράσει ή να παρακάμψει τις δυσκολίες του άρθρου 51 του χάρτη, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία δυνατότητα παράκαμψης ή αποφυγής της εφαρμογής των διατάξεων του χάρτη σε μελιωδών δικαιωμάτων. Τώρα, επόμενη ερώτηση, τι θα γίνει με την άσκηση πλήρων δικαιωμάτων ψήφου ε, στον τόπο κατοικίας. Ε, ακούσαμε διάφορες εναλλακτικές ε, λύσεις, λύσεις μπορούμε να πολεμήσουμε κατά της στέρησης του δικαιώματος, μπορούμε να υποβάλουμε καινούργια μέτρα, μπορούμε να ζητήσουμε τον περαιτέρω συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ε, πολλά σημεία για περαιτέρω συζήτηση. Λοιπόν, η Επίτροπός μου ήδη είναι εδώ και δεν θα ήθελα να την καθυστερήσω και είμαι στη διάθεσή σας ε, για προσωπικές επαφές μετά τη συνέντευξη τύπου. Η κυρία Παπαδοπούλου, θα ήθελα τώρα να, να διακόψουμε, χρειαζόμαστε πέντε λεπτά να τελειώσουμε, αλλά αφού η κυρία Ρέντινγκ... Α, Ωραία. Αφού η κυρία Ρέντινγκ είναι εδώ, θα, να δια... θα πρέπει να διακόψουμε τώρα και διακόπτουμε ώσπου να καθίσει στην έδρα. Thank you all again. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και τη συνεισφορά σας στη ε, σημερινή ημερίδα συζήτησης ε, για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ήγηκε η ώρα τώρα να ακούσουμε τις ε, καταληκτικές παρατηρήσεις από την εξαιρετική μας ομιλήτρια σήμερα το απόγευμα, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ. Ακούσαμε τη σημασία της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, πώς μπορούμε να θεμελιώσουμε την πολιτική συμμετοχή μέσω της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστόματος της κυρίας Ρέντινγκ ε, τι μέλη γενέστε. Κυρία Ρέντινγκ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Αξιότιμα μέλη. Το να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια είναι μια πολύ επίκαιρη ε, επικεφαλίδα ε, και δικαίως επιλέχθηκε για την ακρόαση αυτή, διότι ε, είμαστε στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών και προσεγγίζουμε τα 20 γενέθλια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε τον απολογισμό των όσων έχουμε επιτύχει και να συζητήσουμε τις νέες προπτικές. Προκειμένου να κάνουμε τον απολογισμό, ε, να πούμε ότι το Μάστριχτ δεν ήταν ίσως αυτό το οποίο θα ήλπιζαν πολλοί πριν από 20 χρόνια. Αλλά δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να υποτιμούμε και τι συνέβη πριν από 20 χρόνια, διότι μέσω της δημιουργίας ενός κοινού καθεστώτος για όλους τους Ευρωπαίους και ε, προσδίδοντας αυτό το καθεστώς και μία σειρά από επιπλέον δικαιώματα, τα οποία είναι τόσο θεμελιώδη όσο η ελεύθερη ε, κυκλοφορία και το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε, δόθηκε ένα στεναρό μήνυμα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια αγορά. Είναι κάτι περισσότερο από έναν χώρο ελευθέρου εμπορίου μεταξύ εθνών. Και νομίζω ότι αν το επαναλάβω συνεχώς, ξανά και ξανά και ξανά, μπορεί κάποιοι να εκπλαγούν, διότι ε, ε, φαίνεται, νιώσουν ότι το άκουσαν για πρώτη φορά, αλλά το ακούστηκε για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια. Τότε τέθηκε επιτάπητο στο ζήτημα αυτό και έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύχθηκε σε ένα κοινό χώρο ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους τους τις πολίτες. Διότι πριν από το Μάστριχτ οι Ευρωπαίοι ήταν απλώς οικονομικοί φορείς σε μια ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα. Και 20 χρόνια πριν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννήθηκαν ο Ευρωπαίος πολίτης, ΣΥΤΙΣ Ευρωπαίος ΣΟΥΜ. Αν δεν ήταν άλμα, ήταν τουλάχιστον ένα τεράστιο βήμα προς την πολιτική ολοκλήρωση. Και έκτοτε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει αυτή τη νέα διάσταση επανειλημμένως δηλώνοντας σε αρκετές αποφάσεις ε, από την αρχή της χιλιετίας ότι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια θεωρείται το θεμελιώδες καθεστώς των υπηκών των κρατών μελών. Επαφείται τώρα σε εμά ε, να συνεχίσουμε από αυτό το τεράστιο άλμα και να κάνουμε και μια σειρά από περαιτέρω βήματα προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φρονώ ότι το ευρωπαϊκό έτος αυτό μαζί με την 20η επέτειο ε, και την προετοιμασία των ευρωεκλογών είναι πραγματικά η κατάλληλη στιγμή ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και τι θα πρέπει να σημαίνει το να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις. Δράσεις τις οποίες θα μπορούν να κατανοήσουν οι πολίτες και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα απτά παραδείγματα προκειμένου να επισημάνουμε στους πολίτες ποια δικαιώματα διαθέτουν. Ότι είναι δικαιώματα τα οποία ωφελούν τη ζωή τους, ε, προσφέρουν ευκαιρίες και τα δικαιώματα αυτά αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για αυτά τους τα δικαιώματα. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ. Οι περισσότεροι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρεπιπτόντω σήμερα δημοσιεύθηκε και ευρωβαρόμετρο περί των θεμάτων αυτών, ε, είναι στο διαδίκτυο και εξετάστε το διότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι πολίτε συνειδητοποιούν ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτε, αλλά δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Και νομίζω ότι αποτελεί υποχρέωση να εξηγήσουμε στους πολίτες τι διέπει, τι φέρπει ε, στην ευρωπαϊκή τους ηθαγένεια, στο γεγονός ότι δεν είναι μόνο πολίτες ενός κράτους μέλους, αλλά είναι πολίτες ε, της Υπήρου. Και αυτή ήταν η πρόθεσή μου όταν το 2010 δημοσίευσα την ε, πρώτη έκθεση για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια μαζί με 25 πολύ συγκεκριμένα και εφικτά μέτρα, τα οποία στόχο είχαν να διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωβουλευτές, οι οποίοι και μεμονωμένα αλλά και συλλογικά επεξεργάστηκαν αυτές τις προτάσεις προκειμένου να τις υλοποιήσουν για τους πολίτες. Θα ήθελα εν είδη παραδείγματο να σας πω τι ακριβώς εννοώ με συγκεκριμένα ε, μέτρα και κοντά στη ζωή των πολιτών με μερικά παραδείγματα. Υγεία. Σε γενικές γραμμές οι πολίτες προτιμούν ε, οι υπηρεσίε υγείας να τους παρέχονται κοντά στο σπίτι τους, αυτό είναι λογικό, αλλά ορισμένες φορές υπάρχει ανάγκη για κάποια θεραπεία και οι ασθενεί πρέπει να μεταβούν στο εξωτερικό ή ε, μπορεί το εγκύτερο νοσοκομείο να είναι με, διασχίζοντας τα σύνορα και όχι σε μια κοντινή πόλη στο ίδιο κράτος μέλος. Η οδηγία λοιπόν για την ε, παροχή διαμαθηρεγών υπηρεσιών υγεία, ε, την οποία θα πρέπει να μεταφέρουν τα κράτη-μέλη στο εθνικό του δίκαιο πριν το τέλο του 2013, παρέχει ένα σαφέ πλαίσιο κανόνα για την ε, διασυνοριακή υγεία και δεν θα βελτιώσει μόνο τι δυνατότητε επιλογή, αλλά θα δώσει και την αίσθηση στου πολίτε ότι είναι ευπρόσδεκτοι όταν πηγαίνουν εκτό των συνόρων. Ένα δεύτερο στοιχείο, η προστασία των καταναλωτών. Γνωρίζετε ότι ε, γίνονται κάποιες δράσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε τη σωστή μεταφορά της ε, πιο πρόσφατης οδηγίας για τα ε, δικαιώματα των καταναλωτών πριν από το τέλος του έτους. Τα νέα μέτρα θα ενισχύσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, θα μπορούν να τιμωρούνται αυτοί που διαπράττουν απάτη μέσω διαδικτύου, οι καταναλωτές δεν θα υποχρεούνται να αγοράσουν ανεπιθύμητη ταξιδιωτική ασφάλεια και όλοι θα έχουν 14 μέρες στη διάθεσή τους αν επιθυμούν να επιστρέψουν αγαθά τα οποία αγόρασαν εξ αποστάσεως, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω τηλεφώνου. Προξενική προστασία ε, κατέθεσα μια πρόταση βάσει της οποίας ε, γνωμοδότησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζητάται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Η πρόταση στόχο έχει να βελτιώσει τη συνδρομή των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε περίπτωση κρίσης και κατεπίγουσες περιπτώσεις όταν ταξιδεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαίωμα μη διάκριση στην προξενική προστασία, αυτό νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα από τα βασικά παραδείγματα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και νομίζω ότι μπορεί να παρουσιαστεί και ελπίζω ότι μέχρι τότε θα έχει, ε, θα έχει γίνει εθνικό δίκαιο και θα μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες κατά τις ευρωεκλογές. Ε, και νομίζω ότι σε περιπτώσεις όπως ε, την κρίση της Ιαπωνίας, της Λιβύης και της Συρίας ε, ο ευρωπαϊκός συντονισμός θα διευκρινίσει καλύτερα ποιοι πολίτες μπορούν να περιμένουν και να επωφεληθούν από το τι κάνουν οι προξενικές αρχές. Ελευθερία κυκλοφορίας, θεμελιώδες δικαίωμα. Επειδή από τότε που ανέλαβα το θέμα αυτό, εξετάζω επισταμένα τον τρόπο με τον οποίο έχουν εφαρμοστεί οι οδηγίες ε, από τα κράτη-μέλη. Και ε, θα πρέπει να σας πω ότι με εξέπληξε το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκαν. Ε, έκτοτε βέβαια έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα προς αυτό το σκοπό και πιστεύω ότι πλέον τα περισσότερα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες που περιλαμβάνονται στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία και κάποιοι άλλοι έχουν ε, προσαχθεί στο δικαστήριο. Ενημέρωση προς τους πολίτες. Εδώ και πάλι έχουν γίνει αρκετά για να βελτιωθεί η ενημέρωση προς τους πολίτες, ε, κυρίως μέσω του Europe Direct και του Your Europe, όπου διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και νομίζω ότι αυτό επισημάνθηκε και σήμερα το πρωί. Βέβαια, θα πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα και να μπορέσουμε να αποκομίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Έτο Πολιτών, ώστε να αυξηθούν οι γνώσει των Ευρωπαίων πολιτών για τα συστήματα αυτά τα οποία έχουν στη διάθεσή του. Εξακολουθεί να με σοκάρει το γεγονό ότι ακόμα και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την Ευρώπη δεν γνωρίζουν τίποτα για το Europe Direct ή το Your Europe ε, και την δικτυακή πύλη αυτή. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό οι γνώσεις αυτές ε, να μεταλαμποδευτούν στους πολίτες μας. Αυτά όλα είναι επιτεύγματα. Αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, διότι η ελεύθερη ε, κυκλοφορία και διαβίωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δικαίωμά μας. Και αυτό το δικαίωμα, ε, από ό,τι είδαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο τελευταίο ευρωμαρόμετρο, ε, Εάν οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ένα δικαίωμα, αυτό είναι αυτό το δικαίωμα. Η ελευθερία κυκλοφορίας. Το γνωρίζουν και ξέρουν ότι υπάρχει το δικαίωμα στη μη διάκριση. Γνωρίζουν όμως ότι παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν εξασκούν αυτό το δικαίωμα, κυρίως ε, λόγω ε, υπερβολικής γραφειοκρατίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Ε, κατανοώ ιδιαίτερα επίσης και τις ιδέες ε, που ακούστηκαν από ε, τη, όσα προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση πέρσι. Ε, ξεκίνησε το Μάιο αυτό, είχαμε 12.000 απαντήσεις από πολίτες και μας έδωσαν πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά. Και για παράδειγμα ένας εξ αυτών ζητούσε να βοηθηθεί το προσωπικό, οι υπάλληλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να γνωρίζουν αυτοί τι δικαιώματα έχουν οι πολίτες τους, διότι πολύ συχνά δεν ισχύει. Και βεβαίως ε, πώς μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη οι πολίτες τους τα δικαιώματα όταν η τοπική αυτοδιοίκηση διαθέτει υπαλλήλου που δεν τα γνωρίζει. Και άκουσα και τα δικά σας τα σχόλια για την ε, μείωση του διοικητικού άχθους για τους πολίτες στο μέλλον, ε, κυρίως ε, για έγγραφα τα οποία χρειάζονται όταν μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη. Θα παρουσιάσω στο Κοινοβούλιο περίπου γύρω στο Πάσχα μια συγκεκριμένη πρόταση για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τη χρήση διεθνών, ε, ε, διεθνώς αναγνωρισμένων εγγράφων, πιστοποιητικό γάμου, γεννήσεως και ούτε καθεξής. Και για να είναι σαφές, επειδή ξέρω ότι θα ξανασυμβεί, να ξέρετε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αλλάξει τους κανόνες για το γάμο στα διάφορα κράτη-μέλη. Μην αρχίσετε λοιπόν και πάλι αυτή τη συζήτηση αλλά θα βοηθήσει να πλουστευτεί η ζωή των πολιτών. Ένα έγγραφο είναι ένα έγγραφο και θα πρέπει να αναγνωρίζεται. Και ορισμένες φορές είναι τόσο επαχθείς οι διαδικασίες ε, πιστοποίησης ε, του γνήσιου του εγγράφου ε, οι που θα πρέπει να μειωθούν και θα πρέπει να μειώσουμε τις απαιτήσει ε, πιστοποίησης για μεταφράσεις και αντίγραφα μεταξύ άλλων. Σας παρακαλώ λοιπόν, ζητώ τη συνδρομή σας όταν θα κατατεθεί η πρόταση να την προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερο ώστε να μπορούμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Όσον αφορά τώρα την πρωινή συζήτηση, μπορούμε να εξετάσουμε πιθανές λύσεις όσον αφορούν και άλλα έγγραφα όπως ας πούμε διαμονή, παραμονή, τοποκατοικίας. Υπάρχει λοιπόν, ε, ε, υπάρχουν διαφορετικού τύπου έγγραφα, μια ολόκληρη δέσμη τεκμηρίωσης που μπορούμε να απλουστεύσουμε. Στο ευρωβαρόμετρο 9 από τους 10 Ευρωπαίους πολίτες θεωρούν ότι η ανεργία και η παρούσα οικονομική κρίση είναι η πρώτη προτερότητα, η πιο το πιο κρίσιμο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε ότι όχι μόνο καταπολεμούμε εναντίον της κρίσης, αλλά ότι λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαίτερες ανησυχίες ε, των νέων πολιτών μας ε, για την ανεργία των νέων. Έχουμε γι' αυτό διατυπώσει μέτρα ε, εγγύησης ε, ε, κατάρτισης έτσι ώστε άνεργοι νέοι κάτω των 25 να μπορούν μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες της ανεργίας τους να τύχουν να συμμετάσχουν μάλλον σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης προσόντων. Επίσης έχουμε φροντίσει για την απάλληψη πολλών εμποδίων, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την αναζήτηση εργασίας από τους Ευρωπαίους πολίτες και δι' τους νέους. Παρεπιπτόντας, ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει το εξής Δύο τρίτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει ως αποτέλεσμα οικονομικά ωφέλη. Ωφέλη δηλαδή οικονομικά το κράτος μέλους τους. Και αυτή η ένδειξη θα έλεγα ότι είναι σταθερή και καλύπτει ε, την ευρωπαϊκή επικράτεια. Αυτό σας δείχνει ότι ορισμένες φορές οι πολίτες ε, είναι πιο ρεαλιστές από ότι είναι οι πολιτικοί. Αυτό ως παρένθεση. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα της ελεύθερης διακίνησης θα συνεχίσουν να ε, υπάρχουν, να είναι πολύ ψηλά στην μερίσια διάταξή μας. Και ένα άλλο θέμα που βρίσκεται στην μερίσια διάταξη του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή είναι οι ευρωεκλογέ. Και οι ευρωεκλογέ ε, δείχνουν ότι το πρόβλημα υπάρχει κυρίως στην πάρα πολύ χαμηλή συμμετοχή 43% μόνο Ευρωπαίων πολιτών ψήφισαν σε ευρωεκλογέ. Και ξέρετε τι με ανησυχεί εμένα περισσότερο, ότι στη μεγαλύτερη πλειοψηφία οι μη ψηφίσαντες ήταν νέοι άνθρωποι, νέοι. Ε, ε, ε, ενώ εμείς θέλουμε ειδικά να προσελκύσουμε τους νέους και να τους πείσουμε να ψηφίζουν. Γι' αυτό λοιπόν τον περασμένο Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν την πρότασή μου τη διευκόλυνση της κατάθεσης υποψηφιωτήτων ε, Ευρωπαίων πολιτών ε, για τις ευρωεκλογές και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτό πιστεύω ότι θα φανεί το αποτέλεσμα αυτό στις επόμενες ευρωεκλογές του 2014. Ένα άλλο θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να χειριστούμε είναι τα θέματα των ευρωεκλογών. Συνήθως τα θέματα αυτά ε, είναι, έχουν μια εθνική, έναν εθνικό χαρακτήρα, κρατικό χαρακτήρα. Ενώ εμείς θέλουμε να προβάλλουμε πολύ περισσότερο την ευρωπαϊκή διάσταση, βοηθώντας τους πολίτες να καταλάβουν πολύ περισσότερο τη σχέση μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών διαδικασιών. Παραδείγματο χάρη, πρέπει να τονίσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση ε, των ε, προβλημάτων, να αυξήσουμε την προβολή από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Η Κομισιόν λοιπόν θα υποβάλει περαιτέρω προτάσεις για την ε, εδραίωση της μέγιστης διαφάνειας στις ευρωεκλογές Παραδείγματο χάρη, τι είδου σύνδεσμο έχουν τα ευρωπαϊκά κόμματα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς διαμορφώνεται η εκπροσώπησή τους. Και κοιτάζοντα απευθεία τον κύριο Νταφ, επειδή είναι ειδικό, το άλλο πρόβλημα που μας απασχολεί είναι η στέρηση του δικαιώματος ψήφου. Πράγματι και αυτό το πρόβλημα έχει μια πολύ ε, έχει μια πολύ σημαντική ε, θέση στην ατζέντα μου και έχουμε αποφασίσει ότι θα αφιερώσουμε μια συνεδρίαση ε, σε αυτή τη συζήτηση αποκλειστικά αυτού του θέματος. Έχουμε λοιπόν τώρα ε, καθήκον να σκεφτούμε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, να αναλογιστούμε αυτά που είπατε και να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις. Λοιπόν, στο θέμα των λύσεων, η έκθεση για τους Ευρωπαίους πολίτες θα παρουσιαστεί θα, κατά τις 9 Μαΐου φέτος. Και πάλι εδώ θα δείτε ότι θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένες δράσεις για πρακτική εφαρμογή. Αλλά ο στόχος μας κυρίως είναι να αυξήσουμε την γνώση, τη συνειδητοποίηση. Αυτή η Ευρώπη του μέλλοντος που θέλουμε να οικοδομήσουμε και που θα οικοδομήσουμε θα βασιστεί σε μια πολιτική ένωση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη. of if the are Και όλα αυτά και οι ευγενείς στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν ε, αν δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή διάσταση. Πέραν της, Ευρωπα... της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης πρέπει να ασπαστούν οι πολίτες μας στο αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Γι' αυτό ακριβώς ανακουφίστηκα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου που έδειξαν ότι η τεράστια πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών αισθάνονται Ευρωπαίοι αυτό λοιπόν είναι πολύ καλό σημείο εκκίνησης. Και αυτό ισχύει για τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Αλλά, εκτός από την ελεύθερη κυκλοφορία, έχουμε διαπιστώσει ότι οι πολίτες μας δεν γνωρίζουν ούτε τα δικαιώματα, ούτε τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό πρέπει να αλλάξει και η αλλαγή αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Πρώτον, με, την, με το έτος αυτό ε, ως, ευρωπαϊκό, ως έτος του Ευρωπαϊκού Πολίτη. Θα δείτε και άλλα σημάδια με, στην διαμόρφωση της, ε, των, της για, τους, ε, για την ευρωεκλογή, τις ευρωεκλογές και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτό θα φανεί του χρόνου στις εκλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ για την ε, ε, παρουσίασή σας και σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα προγράμματα, τα, όλο αυτό το εμπεριστατωμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών που παρουσιάσετε, τι πρέπει να γίνει, τι θα κάνετε και τι λύσεις, σε τι λύσεις στοχεύετε. Εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας και στο μέλλον. Σας είμαστε πάντοτε στην, στο πλευρό σας να σας στηρίξουμε, παρόλο που έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Έχουμε τώρα την συνέντευξη τύπου μια άλλη αίθουσα. Και θα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 If I may have your uh, attention, please, we would like to ask Mrs. Adamo to come. Ελάτε παρακαλώ στο πάνελ, η κυρία Άνταμο και οι τελευταίες δύο μιλήτε, για να μπορούμε να, για να μπορέσουμε να τους ακούσουμε. Δεκαπέντε λεπτά για τις ερωταπαντήσεις στους τρεις τελευταίους, ε, στα τρία τελευταία μέλη του πάνελ.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 So I like to give the floor to Mrs. Eh, Catherine ε, Θα ήθελα λοιπόν να ε, επανέλθουμε στην κυρία Κεσεντζιάν. Δύο λεπτά για να ολοκληρώσει. Μετά ο κύριο Σουμπιώτο να ολοκληρώσει. Και αν υπάρχει διάθεση άλλων ερωτήσεων, ε, θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε. Κυρία Πρόεδρε, οι ερωτήσεις που γίνανε, βλέπω όμως ότι φεύγει το μέλος που κάνει μια ερώτηση. Το θέμα την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις χώρες μέλη, αν λειτουργεί καλά, αν κάνει τη δουλειά του. Προσωπικά θα πω ότι δεν έχω ιδέα. Ξέρω που είναι τα κτίρια, που είναι τα γραφεία της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στο Παρίσι, αλλά ειλικρινά δεν έχω ιδέα το τι κάνουν, δεν είχα καμιά επαφή με αυτούς, δεν ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Δεν θυμάμαι να είχα, και όταν χρειάστηκε, δεν θυμάμαι να είχα μια ουσιαστική βοήθεια. Ε, με ενοχλεί κάπως, σαν είχα, μήχανα, αλλά αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να δώσω. Ε, για το άρθρο 51 της χάρτας τώρα ε, ειλικρινά εκπλήσουμε που θέτει κανείς και την ερώτηση. Δεν μπορεί πάει να πάει ενάντια κανείς στον κατα... στη διάκριση των εξουσιών. Αυτό υπάρχει στο δικαίωμα, το ευρωπαϊκό δίκαιο, στις συνθήκες, εκτός κι αν ξαναλάξει κανείς στις συνθήκες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, έχουν κουραστεί να μην υπάρχει κάποια σταθερότητα, κάποιες σταθερές. Όλη την ώρα όλα αλλάζουν. Αυτό οδηγεί σε μια πίθανη κατάσταση και δεν μπορεί κανείς να ξέρει τα δικαιώματά του. Έχουμε την ε, διάκριση του εξουσιών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μέλη. Δεν μπορεί κανείς να πάει ενάντια σε αυτά, σε αυτές εξουσίες. Αλλά, όπως και είπα σήμερα το πρωί και νομίζω είναι σημαντικό, θα μπορέσει κανείς να δουλέψει στο να έχει μια καλύτερη εφαρμογή αυτό που λέμε best practice, λέω τον αγγλικό όρο. Ε, στα, γιατί στα, άμα πούμε τις βέλτιστες πρακτικές στα γαλλικά τέλος πάντων δεν σημαίνει τίποτα. Επίσης το benchmark που λένε στα αγγλικά. Αυτό είναι σημαντικό θα πρέπει να έχουμε τα καλύτερα τα παραδείγματα σε κάποιες χώρες όσον αφορά την διοίκηση και με αυτόν τον τρόπο να πείσουμε και τις άλλες χώρες μέλη. Δηλαδή ξανά ερχόμαστε στο θέμα που έχει να κάνει με την παιδεία, κατάρτιση. Ε, αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κεσεριάν. Κύριε Σουμπιώτο, έχετε το λόγο. Δύο σχόλια έχω να κάνω. Πρώτον, για αυτά τα οποία ακούσαμε από την παρέμβαση του κυρίου Χέφνερ, ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε να εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, από τους εκπροσώπους του λαού, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος ε, ο οποίος εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά ε, όργανα θα πρέπει να είναι ερετός κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο. Και εδώ δεν μιλώ ως νομικός, ως δικηγόρος, μιλώ ως Ευρωπαίος πολίτες. Είναι απαράδεκτο. Το παράδειγμα το οποίο έρχεται στο νου είναι η δημιουργία μιας κοινή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση από τα κράτη-μέλη, ε, αντί να εκπροσωπείται το πρόσωπο τη Ευρώπη στο διεθνέ ε, προσκήνιο, ήταν σαφές ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, ήθελαν να ε, μειωθούν τα εθνικά τους δικαιώματα από την εξωτερική υπηρεσία δράσης και ε, διόρισαν έναν άνθρωπο που δεν είναι τόσο χαρισματικός επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας, τη λέει Κάθριν Άστον. Αν λοιπόν θέλετε πραγματικά να δημιουργήσετε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, θα πρέπει να υποστηρίζετε τι συνέπειε και να ψηφίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτε κάποια προσωπικότητα, η οποία θα είναι σε θέση να είναι η φωνή τη Ευρώπη ε, στο διεθνέ προσκήνιο. Ένα σχόλιο είναι αυτό. Το δεύτερο σχόλιο μου είναι ότι με αποθάρρυνε λίγο η παρέμβαση του κυρίου Νταφ υπό την έννοια ότι ε, είχε την ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσυπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επομένως το άρθρο 3 της Σύμβασης κατά κάποιο τρόπο θα αποτελέσει τη λύση στα προβλήματά σας στα προβλήματά μας. Ε, είπα όμως στην παρέμβασή μου ότι έχουμε πάνω από 40 χρόνια συστηματικής νομολογίας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μεταφράζει το άρθρο 3 της σύμβασης που λέει ότι δεν ε, παραβιάζεται κανένας εθνικός νόμος που στερεί το δικαίωμα ψήφου ατόμων που διαμένουν ε, εκτός της χώρας τους. Αυτό γίνεται κατ' επανάληψη, κατά συρροή, είναι από το 1976. Το να θεωρεί λοιπόν κάποιο ότι η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το άρθρο 3 θα αλλάξει τα πράγματα, είναι φρούδες ελπίδες. Το 1964 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε και ε, ότι υπάρχει ένα σύστημα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πρέπει να έχει δικό του σύστημα. Δεν χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι κανόνες στη συνθήκη αρκούν για να εγγυηθούν στους Ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές ακόμα και αν διαμένουν εκτός της χώρας τους. Τελεία. Δυστυχώ, ο κύριος Νταφ που έθεσε την ερώτηση δεν είναι εδώ, θα μπορούσε να σας απαντήσει. Και για να είμαστε δίκαιοι με όλους, εάν υπάρχει κάποιος που δεν είχε την ευκαιρία να ρωτήσει κάτι και θέλει, παρακαλώ αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, απλώς ε, θέλετε συστηθείτε μας. Τρεις, ωραία. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τον κύριο απέναντι με τον κύριο απέντη μου. Παρακαλώ πείτε το όνομά σας. Α, το όνομά μου είναι Φιλίπ. Εγώ είμαι 38 ετών, γεννήθηκα στην Ιταλία, έζησα στη Γαλλία και στην Ελβετία και κατέληξα στο Λονδίνο. Εάν θέλετε συμμετοχή, θα πρέπει να μας αποδείξετε ότι η συμμετοχή μας δημιουργεί μια συγκεκριμένη, έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Ε, εάν θέλω να σας θυμίσω να κάνω έναν παραλληλισμό με το κινέζικο πολύμπυρο όπου 26 μέλη εκλέξανε τον πρόεδρο του κινέζικου πολύμπυρο ο οποίος ε, ε κυβερνά ε, ένα μισή δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο κύριος Μπαρός εκλέχθηκε από 27 από το κολέγιο των επιτρόπων. Λοιπόν, ε, εάν θέλετε και το λέτε ειλικρινά να συμμετάσχουν οι νέοι και να ψηφίσουν, πρέπει να αλλάξετε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας αυτού του σώματος και να μας αποδείξετε ότι δεν είμαστε παθητικοί συμμετέχοντες, αλλά είμαστε δραστήρια ενεργά μέλη. Και εφόσον θέλετε τη συμμετοχή μας, πρέπει να δούμε και εμείς τα απτά αποτελέσματα. Είδατε με το θαυμάσιο παράδειγμα της Wikipedia πώς μπορεί συλλογικά και παγκόσμια ο πολίτης να συμμετάσχει στη διαμόρφωση μιας εγκυκλοπαίδειας. Λοιπόν, παραδείγματα υπάρχουν. Εάν θέλετε ευρωπαϊκή συμμετοχή, χρειάζεται μια αναθεωρημένη, μια νέα κοινωνική ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ το όνομά σας. Δεν άκουσα το όνομά σας, λέει η πρόεδρος. Η πρόεδρος ζητάει το όνομά του να το γράψουμε. Φιλίπ Πατάρη. Ε, ευχαριστώ πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία.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 και είμαι και ιδρυτικό μέλος της πρώην ε, Ένωσης για τα Δικαιώματα των Βρετανών στο εξωτερικό και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σουμπιώτο και την ε, κυρία Κότρο για την ε, μακροσκελή και πολύ εύστοχη επεξήγηση της κατάστασης των Βρετανών που διαμένουν στο εξωτερικό και του δικαιώματος ψήφου τους. Ε, υπήρξαν κάποιες εξελίξεις. η Βουλή των Λόρδων τον Ιανουάριο ανέφερε ότι θα συσταθεί ε, μια νέα διακομματική επιτροπή για να εξετάσει το θέμα των δικαιωμάτων ψήφου για τους ε, Βρετανούς ε, ψήφου, ψηφοφόρους στο εξωτερικό ευρύτερα και φαντάζομαι ότι στη συνέχεια θα περάσει και από την Βουλή των Κοινοτήτων και από τη Βουλή των Λόρδων. Το θέμα όμως είναι πιο περίπλοκο διότι εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να ψηφίσουν ακόμα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανάλογα με τη φύση λοιπόν της ε, ε, σχέσεις που έχουν με τη χώρα τους οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορεί να μπορούν ή να μην μπορούν να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογέ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, είναι μια πολύ ουσιαστική έλλειψη, διότι περίπου 35 με 60 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν μπορούν να ψηφίσουν. Και δεν ισχύει μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, φυσικά, και, αλλά και για τους Έλληνες που δεν έχουν πάντα την δυνατότητα να ε, μεταβούν να ψηφίσουν, διότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει σε ε, πρακτικό δίκαιο τμήμα του συντάγματός της. Ε, το ίδιο ισχύει και για την Ιρλανδία, τη Μάλτα, τη Δανία και αν δεν κάνω λάθος και για την Κύπρο. Ε, όπως ε, άκουσα νωρίτερα και μάλλον είναι και άλλες οι χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να επεκτείνει το δικαίωμα ψήφου το πρακτικό δικαίωμα ψήφου για τις ευρωεκλογέ, ε, αν όχι και για τις εθνικές εκλογές, ε, πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Κάποιοι, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή του να υπάρχει μια συνεχής ψήφος για τη χώρα τους ή μια ψήφος ε, για τη χώρα διαμονής τους, λένε συνήθως ότι θα πρέπει να επιλέξω ένα εκ των δύο. Γιατί να επιλέξουμε, αν έχει κάποιο ένομα δικαίωμα να ψηφίζει είτε στη μία είτε στην άλλη χώρα και στις δύο, γιατί να μην ψηφίζει και στις δύο. Αν κάποιος έχει διπλή υπηκότητα, διπλή ε, υπηκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην μπορεί να ψηφίσει και σε κάθε μία από τις χώρες του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Και τελευταίος ομιλητής ο κύριος ε, Γκλυξιών. Εξ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι μέλος ε, της πρωτοβουλίας ε, για το δικαίωμα ψήφου και στόχος μας είναι να υπάρχει δικαίωμα ψήφου για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στη χώρα τους. Είναι λίγο διαφορετικός τρόπος ρύθμισης του προβλήματος το οποίο ε, επικαλεστήκατε προηγουμένως ε, και αφορά μόνο τους Βρετανούς. Η κυρία Κοτιλέρ, Κοντερίλ, συγγνώμη, ε, έκανε έκκληση την οποία δεν θα επαναλάβω Δύο παρατηρήσεις και μία ερώτηση από πλευράς μου. Καταρχάς, η παρατήρηση είναι ότι μία απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς αυτό το σκοπό για το δικαίωμα ψήφου μπορεί να ληφθεί επί τη βάση της ε, κείμενης συνθήκης. Έχουμε το άρθρο 27 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Νταφ. Η διαδικασία είναι μακρά, αλλά υπάρχει. Το Συμβούλιο μπορεί να διευρύνει τον κατάλογο των δικαιωμάτων που καθορίζονται στη συνθήκη. Πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζήτηση από το Συμβούλιο, ομοφωνία των κρατών μελών, κύρωση από κάθε κράτο μέλο. Η διαδικασία είναι μακρά, αλλά ε, τουλάχιστον με πολιτική βούληση είναι δυνατή. Δεύτερον, θα ήθελα να σας καταθέσω τη μαρτυρία μου για την πρωτοβουλία Let Me Vote για να σας πω ότι, και δεν θα πω και τίποτα πρωτότυπο, διότι έχουν γίνει ιδιαίτερα σεμινάρια που ε, είναι αφιερωμένα στον κανονισμό αυτό, έχουμε ιδιαίτερες δυσκολίες να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτά τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε, και νομίζω ότι αυτό απουσιάζει από τον κανονισμό, μία νομική βάση η οποία πραγματικά επιτρέπει να βοηθήσουμε συγκεκριμένα την ε, κοινωνία των πολιτών. Υπάρχει η δυσκολία του προϋπολογισμού. Ε, αυτό το γνωρίζουν όλοι. Υπάρχουν ε, δυσκολίες από πλευράς πληροφορικής για τη δημιουργία των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία θα μας επιτρέπουν να κάνουμε συλλογή των στοιχείων online και θα έπρεπε να μας ε, ε δανείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σέρβες της στο Λουξεμβούργο για να υπερβούμε τα προβλήματα σε πρώτο επίπεδο. Και υπάρχει και θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, διότι όπως προβλέπεται το καθεστώς στον κανονισμό δεν επαρκεί, ε, διότι δεν είναι ακριβές. Γίνεται συλλογή σε 27 κράτη-μέλη ποιος είναι ο εθνικός νόμος που εφαρμόζεται για αυτή τη συλλογή δεδομένων. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός νόμος και όχι να εφαρμόζονται 27 διαφορετικοί νόμοι για να υπάρχουν 27 διαφορετικές δηλώσεις για κάθε μία από τις 27 εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των δεδομένων. Ποιο είναι ο εθνικό νόμο, λοιπόν που ισχύει σε αυτή την περίπτωση, εμεί δεν γνωρίζουμε. Ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει. Περιμένουμε λοιπόν την απάντησή τους. Και μια τέταρτη δυσκολία, η οποία είναι πιο σημαντική για μας, διότι η πρωτοβουλία μας ε, απευθύνεται όχι μόνο αποκλειστικά, αλλά ιδίω στους πολίτες που ζουν σε χώρα άλλη ε, της καταγωγής τους, ε, τις οποίες διαθέτουν την ηθαγένεια επειδή ακριβώς είναι πολύ σύνθετα τα πράγματα και τίθενται όρια από τα κράτη-μέλη. Τίθενται λοιπόν αυτοί οι όρια από τα κράτη-μέλη για τη συλλογή των υπογραφών. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ε, ταυτοποίησης, για παράδειγμα μια ταυτότητα ή ένα διαφατήριο. Ε, ή θα πρέπει απλώς να γίνονται δεκτές οι υπογραφές των κατοίκων και μόνο. Και θα ολοκληρώσω σε 30 δευτερόλεπτα διαπιστώνεται ότι κάποιοι πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες, που διαμένουν σε χώρα που δεν είναι η χώρα καταγωγής τους, απλώς και μόνον αποκλείονται από τη διαδικασία. Η κυρία Κότεριλ έφυγε, αλλά εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση. Πρόκειται για Βρετανίδα υπήκαιο, η οποία διαμένει στην Ισπανία και δεν μπορεί να υπογράψει την πρωτοβουλία Let Me Vote. Είναι παράδοξο αυτό, ε, και αυτό είναι απλώ και μόνο ένα παράδειγμα, υπάρχουν και άλλα, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, προκειμένου να υπογράψει κάποιο, ε, προβλέπει ότι πρέπει κάποιο να είναι κάτοικο. Ενώ στην Ισπανία, στην οποία διαμένει η κυρία, για να υπογράψει, θα πρέπει στον υπολογιστή του κάποιο να συμπεριλάβει είτε τον αριθμό τη εθνική του ταυτότητα, είτε τον αριθμό του διαβατηρίου του. Και μία ερώτηση λοιπόν προς τον κύριο Σουμπιώτο. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Γιατί σας έδωσα πολύ χρόνο. Κάνετε πολλά σχόλια. Η κυρία Κεσεντζιάν πρέπει να φύγει. Λοιπόν, τη δίνει τη λόγο να απαντήσει. Ο κύριος Σουμπότο, Σουμπιώτο και η κυρία Άνταμο θα είναι οι τελευταίοι μιλητές. Κυρία Κεσεντζιάν. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που θα πρέπει να φύγω. Τώρα, σε σχέση με την ψηφοφορία, εκπλήσουμε που ακούμε Ευρωπαίοι πολίτες ε, λένε μπορούν να ψηφίσουν για τις ίδιες ε, εξ, εκλογές, ε, δεν ψηφίσουν διπλά για τις ίδιες εκλογές. Αυτό δεν είναι ηθικά σωστό. Ο υπάρχει χώρα καταγωγής ή χώρα υποδοχές, ότι μπορεί να κάνει μια τέτοια εκλογή είναι λογικό. Αλλά το να ψηφίσει κανείς διπλούν δεν μου φαίνεται και σωστό. Ε, όλα στρέφονται γύρω από τη, για τη δημασία της, του τόπου διαμονής σε σχέση με την υπηκότητα. Δεν πρέπει κανείς να αμφισβητεί αυτό που λέει η συνθήκη, δηλαδή ότι η εθνική ε, η εθνικότητα ενός χώρου μέλους είναι αυτή που οδηγεί στην ευρωπαϊκή θαγένεια. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Αλλά θα μείνουμε με το δίκαιο το οποίο ισχύει. Αν δέχεται κανείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια είσοδος για την ηθαγένεια η οποία θα είναι διαφορετική, οδηγούμε σε μια άλλη σειρά προβλημάτων. Ακόμα και αν συμφωνώ με τον εξαριστερόν ε, συνάδελφο, διότι υπάρχει πάντοτε ε, το θέμα συζήτηση πόσες, πόσα χρόνια κτλ. θα πρέπει κανείς να, είναι, ε, να διαμένει σε ένα τόπο. Υπάρχει φυσικά μετά το θέμα της συνηθισμένου τόπου διαμονής, υπάρχει ένας κανόνας πανευρωπαϊκός, ο οποίος ισχύει για όλους, για όλες τις χώρες μέλη, που επιτρέπει κάποιον την άσκηση των δικαιωμάτων. Μπορεί να πει κανείς ότι η διαμονή, ε, έξι μηνών λοιπά, Όλα αυτά μπορεί να συζητηθούν. Ε, αλλά για μένα αυτά τα πράγματα μάλλον είναι σχετικά εύκολα για, να συγκλίνουμε κάπου. Διαυκρίνηση ζητάει ο μιλητής. Θα είμαι τηλεγραφικός. Θα μίλησα πολύ γρήγορα, γιατί προφανώς δεν, δεν με καταλάβατε όταν εννοούσα. Δεν εννοούσα ότι ε, πολίτες που έχουν δύο υπηκό, διπλή υπηκότητα ψηφίζουν δύο, δύο φορές. Όχι. Ε, έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ στη χώρα καταγωγής τους ή μία από τη χώρα τέλος πάντων που τους αφορά, δηλαδή καταγωγής ή διαμονή τότε θα ψηφίσουν μία φορά. Ε, στο κοινοβούλιο μπορεί κανείς να ε, ψηφίσει συνήθως ε, στη χώρα διαμονής του. Τώρα, αν έχω διπλή υπηκότητα, ας πούμε Βρετανική και Δανέζικη, Κάθε χώρα μπορεί, κάθε μία από τις δύο αυτές χώρες μπορεί να πάρει αποφάσεις που επηρεάζουν βασίτατα εμένα και την οικογένειά μου. Γι' αυτό ας πούμε ότι εγώ αποφασίζω θέλω επισημό να ψηφίζω ή στη Δανία ή στη Βρετανία, ανάλογα που βρίσκουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να, να βασίζουμε το θεμελιώδη δικαίωμα, δικαίωμα του της ψήφου μόνο στη διπλή υπηκότητα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και ο κύριος Σουμπιώτο τώρα και συμφωνώ, λέει ο κύριος Σουμπιώτο, ότι βεβαίως υπάρχει ένα θεμητό επιχείρημα να ψηφίζει κανείς ε, και στις δύο χώρες αλλά θα έλεγα να μην είμαστε υπερβολικά φιλόδεξοι, ας κατοχυρώσουμε καταρχάς το δικαίωμα της ψήφου μία φορά, άπαξ και μετά βλέπουμε τι θα γίνει για περισσότερες φορές. Ε, το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να παραβιάζονται διατάξεις του νόμου είτε στο γερμανικό είτε στο γαλλικό δίκαιο. Εάν έχεις διπλή υπηκότητα, ορισμένες χώρες υποχρεώνουν να διαλέξεις την υπηκότητά σου και πού θα ψηφίζεις. Ο γαλλικός νόμος απαιτεί στα 18. Ή έχω τέσσερα παιδιά, δεν θα μπορούσαν, έχουν το δικαίωμα να έχουν διπλή υπηκότητα, αλλά δεν θα το κάνουν δυο λόγου του νόμου. Πρέπει να επιλέξουν. Δυστυχώς δεν κατάλαβα την ερώτησή σας, ε, αλλά νομίζω ότι μάλλον ήρθατε ε, θέμα την ευκολία εγγραφής όταν κάποιος ε, μένει σε μια χώρα που δημιουργεί πρόβλημα. Η ερώτηση μου αφορούσε την κατάσταση, η οποία απορρέει από τον κανονισμό. διαπιστώνουμε ότι κάποιοι πολίτες που διαμένουν σε μια χώρα που δεν είναι η χώρα καταγωγής τους, όπως η περίπτωση της κυρίας Κοτερίλ που ε, Βρετανίδα που διαμένει στην Ισπανία, η συγκεκριμένη δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει. Ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι κάποιο μόνιμος κάτοικος για να ψηφίσει, ε, για να εγγραφεί, συγγνώμη και να υπογράψει, ε, ούτε στην Ισπανία, διότι για να εγγραφεί ε, θα πρέπει να έχει τον αριθμό ισπανικής ταυτότητάς της ή τον αριθμό του ισπανικού της διαματηρίου Και η ερώτησή μου είναι αν κατά την άποψή σας αυτό αποτελεί παραβίαση θεμελιώδης δικαιώματο. Για να μπορέσει να ψηφίσει κάποιο στις τοπικές εκλογές ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι. Για να μπορεί να υπογράψει την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν έχω κάποια αρμοδιότητα επί του ζητήματος. Ε, λυπάμαι. Η κυρία Άνταμο ε, θα μας καλύψει όλους. Έχει όλες τις απαντήσεις. Λοιπόν, θα απαντήσω σε μερικά ερωτήματα. Στον εκπρόσωπο των νέων φεντεραλιστών με εκπλήττει το γεγονός ότι μπορέσετε στις ευρωεκλογέ μιλάμε δύο φορές Εν πάση περιπτώσει λέει ομιλείται η κυρία Ανταμό ότι υπάρχει μία διάταξη που δεν επιτρέπει τη διπλή ψηφοφορία στις ευρωεκλογέ. Ακριβώς λοιπόν για να αποφύγουμε αυτό έχουμε ένα μηχανισμό που υπάρχει στην οδηγία 9301 για να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις. Όπως είπε και η Επίτροπος, θα εκδώσει η Κομισιόν ανακοίνωση σύντομα, σε ερχόμενους ένα-δύο μήνες, που θα διευκρινίζει ακριβώς πώς θα μπορούν οι, ε, τα διοικητικά όργανα των κρατών μελών να ενεργούν πιο αποτελεσματικά χωρίς να υπάρχουν παραθυράκια και κενά. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου για να την αποφυγή της διπλής ε, ψήφου. Τώρα, ε, όσον αφορά την εθνική εισαγένεια σε διάσταση με την ευρωπαϊκή εισαγένεια αυτή τη στιγμή έτσι όπως ορίζουν οι συνθήκες το άρθρο 20 λέει ότι η εισαγένεια της η ευρωπαϊκή δεν αντικαθιστά την υπηκότητα δεν αντικαθιστά την ε, εθνικότητα ενός πολίτη που ανήκει σε ένα κράτος μέλος, έχει την υπηκότητα του κράτους μέλους με τα δικαιώματα του κράτους μέλους αυτού. Τώρα, ε, αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση για υπηκόους τρίτων χωρών, αυτό είναι άλλο θέμα. Η Κομισιόν ήδη στην ατζέντα της για ενσωμάτωση ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την πολιτική συμμετοχή και να ενθαρρύνουν πολίτες να, να ψηφίζουν τοπικά και στις τοπικές ε, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Πιστεύω ότι ε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη νομική βάση να προχωρήσουμε πέραν αυτού. Η Κομισιόν όμως έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλει να ενισχύσει και να διευρύνει ακόμα περισσότερο αυτή την ενσωμάτωση. Όσον αφορά τώρα τον εκπρόσωπο της Ένωσης, η Ευρώπη σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν πράγματι πολλοί απόδημοι Ευρωπαίοι και το ξέρουμε αυτό και τα προβλήματά τους. Είναι ένα θέμα το οποίο ρυθμίζεται από τα κράτη-μέλη. Ορισμένα επιτρέπουν στους πολίτες τους να ψηφίσουν ε, στο εξωτερικό, αλλά δεν επιτρέπουν Τώρα τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις διαφορές και τα διαφορετικά καθοστώτα. Εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ε, χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας ε, για να μπορέσουν να διευκολύνουν τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε ψηφός εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικά. Έτσι θα ενισχύσουμε και τη συμμετοχή. Και η τελευταία παρατήρηση του κύριου Μπραν. Για το άρθρο 25. Πρέπει να προσθέσουμε μέσα στο πλαίσιο συζήτησης για την αποφυγή στέρησης δικαιωμάτων ψήφου και το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές από πολιτών. Σας, ε, σας είπα ότι η Κομισιό προσπαθεί να βοηθήσει όταν ζητάτε η παροχή συμβουλών στην ε, πληροφορική, ε, στις, στις ηλεκτρονικές διαδικασίες και βεβαίως γνωρίζουμε στην αρχική μας πρόταση για το κανονισμό. Γνωρίζουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών έτσι, και ζητούμε ακριβώς την εδραίωση ομοιόμορφων διατάξεων και η τελική έκδοση του κανονισμού είχε ζητήσει διαφορετικές διαδικασίες. Δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε τις διαφορετικές διαδικασίες, διότι ορισμένα κράτη-μέλη ζητούσαν τη συλλογή διαφορετικών στοιχείων και αναγκάσαμε να κατεβάσουμε τον πύχη. Και μια τελευταία παρέμβαση. Είμαι ο πρόεδρος αυτής της Ένωσης Europeans Throughout the World. Ε, Παπαχριστόπουλος λέγομαι. Και θα ήθελα τώρα να, να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Όταν μιλάμε ε, τη, τα δικαιώματα διαμονής και τόπος διαμονής πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κινητικότητα. Πέντε χρόνια στη Γερμανία, τρία στη Δανία, δύο στην Αγγλία. Ε, το θέμα είναι ότι αυτός ο μετακινούμενος πολίτης θα ψηφίσει στη χώρα καταγωγής του. Διαφορετικά θα αναγκαστεί να ψηφίζει σε τρεις χώρες με μια πολύ επιβαρημένη διαδικασία. Και, το, και κάτι άλλο ε, που με εντυπωσίασε είναι ότι είχαμε τόσους πολλούς νέους συμμετέχοντες. Πλειοψηφία θα έλεγα ήταν νέοι και έχουμε μια νέα κατάσταση μετανάστευση στην Ευρώπη, εσωτερική μετανάστευση ανθρώπων νέων που από τις νότιες χώρες μετακινούνται προς ε, βόρειες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι αυτό ε, βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όχι μόνο διότι έχουμε μία ε, στέρηση ε, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, δηλαδή ε, μικραίνει δεξαμηνή εγκεφάλων και ικανών που έχουμε στην Ευρώπη, αλλά θα έχουμε και αυξημένα προβλήματα Ευρωπαίων πολιτών που μεταναστεύουν. Θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ. Κύριε Αντάμου, δύο είναι τα θέματα σε αυτή την περίπτωση. Καταρχάς, θεωρούμε ότι κάποιος θα πρέπει να έχει δικαίωμα ψήφου στη χώρα καταγωγής του και όχι να, την αποκτή, να το αποκτήσει στη χώρα διαμονής του. Και από εκεί και πρέπει επισημάνεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα των νέων ε, και το πώς ε, επηρεάζει αυτό τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η κυρία Κότεριλ, η συντάκτρια της αναφοράς, ανέφερε τις κόρες της. Οι τρεις νέες κόρες της κυρίας Κότεριλ είπαν ότι επειδή ούτως ή άλλως μένουν στην Ισπανία εδώ και αρκετά χρόνια, ούτω η, εμπειρία ψήφου τους εκεί και όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς δεν υποστηρίζουμε αυτή τη μορφή του εκλέγην και του εκλέγεστε, αλλά να πω ότι το θέμα δεν είναι τόσο εύκολο και ίσως θα μπορούσε να γίνει μια πιο διεξοδική συζήτηση να τεθεί το ερώτημα κατά πόσον ο πελίτη θα πρέπει να έχει δικαίωμα να επιλέξει, αν θα πρέπει να δημιουργήσουμε την νομοθεσία γύρω από το δικαίωμα επιλογή του πολίτη ή όχι, ε, ή αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα των τοπικών εκλογών που μπορεί κάποιο να ψηφίσει δύο φορέ σε δύο διαφορετικέ χώρε ή το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου δεν θα μπορεί κανεί να διπλοψηφίσει. Ε, διότι στο τέλος η ψήφος θα σημαίνει ότι θα έχετε δύο ψήφους στο Συμβούλιο Υπουργών. Ε, Υπάρχουν ε, λοιπόν ερωτήσεις ε, με το τι γίνεται με τη στέρηση του δικαιώματος ψήφους, αλλά νομίζω ότι ε, σήμερα ήταν μια πολύ χρήσιμη μέρα και μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ωραία. Με αυτό νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ε, ευχαριστώ ιδιαίτερα τους ομιλητές, ε, τους συμμετέχοντες, τη γραμματεία και τους διερμηνείς ευχαριστή πρόεδρος. Ευχαριστούμε και εμείς και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και τη συμμετοχή σας.